Uh, Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, παρακαλώ καθίστε αν βρείτε κάθισμα. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους στη δημόσια ακρόασή μας για τη χορήγηση των εκχωρήσεων. Υπάρχει ο εισηγητής μας, που οργανώνει την ακρόαση και καλωσορίζω και τους εμπειρογνώμονες Επίσης πολλοί παρίστανται εδώ ως κοινό. Η αίθουσα αυτή βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα έπρεπε, αλλά να. Επίσης καλωσορίζω όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Πρέπει να ξέρουν λοιπόν οι εμπειρογνώμονες ότι θα καταγραφούν οι παρεμβάσεις τους για την αιωνιότητα. Έχουμε και άλλη αίθουσα χωριστή ακροάσεως που ακούγεται, που ακούγονται οι παρεμβάσεις. Για να δω ποιοι έχουν γνωμοδότηση. Υπάρχει και η έκθεσή μας. Υπάρχουν άλλες επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν για μας. Νομική Επιτροπή Βιομηχανίας και Διεθνούς Εμπορίου και Απασχόλησης. Ωραία. Στους φακέλους σας πρέπει να έχετε ένα αντίγραφο των βιογραφικών, των εντυπωσιακών βιογραφικών των εμπειρογνωμόνων μας. Ο καθένας θα έχει δέκα λεπιτά. Πρώτος γύρος. Καθορισμός του εργαλείου. Δεύτερος γύρος τι είδους καθεστώς θέλουμε. Ελαφρό λέει καθεστώς ο τίτλος. Ο εισηγητής μας τα καθόρισε αυτά. Τον καλό λοιπόν να μας εκφράσει τις βασικές του σκέψεις και μετά θα αρχίσει ο γύρος των εμπειρογνωμόνων. Ο κύριος Φίλιππος Ζουβέν λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζω. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καλέσουμε όλους όσους θα ήθελαν να συμμετέχουν στην εκδήλωση. Αυτή χρειάστηκε μια επιλογή μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. Υπάρχουν και οι σκιώδεις που είχαν την καλοσύνη να προσέλθουν μεταξύ των οποίων και η κυρία Ρούλα. Το κείμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι οι εκχωρήσεις είναι θέμα πολύπλοκο και που παίρνει πολλές μορφές, πολύμορφο. Ακόμη και μόνο γι' αυτό δικαιολογούνταν οι Υπάρχει και σοβαρή νομολογία που μας δείχνει ότι πρέπει να υπάρχουν συντονισμένοι, συνδυασμένοι κανόνες για τις εκχωρήσεις. Ορισμένοι θα ήθελαν το κείμενο αυτό να είναι πολύ πιο δεσμευτικό, άλλοι πολύ λιγότερο, δύσκολη η πολιτική, σαν την καλογερική και ελπίζουμε η σημερινή ακρόαση να μας φωτίσει ορισμένες τουλάχιστον πτυχές του προβλήματος για να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ Φιλίπ για την σαφή αυτή παρουσίαση. Φυσικά θα λάβει το λόγο και στο τέλος της ε, ακρόασης. Προχωράμε τώρα στο πρώτο ομιλητή μας τον κύριο Μπερνέτ, ο οποίο είναι ειδικό στα λογιστικά θέματα και έχει πολλαπλή εμπειρία σαν σύμβουλο επιχειρήσεων για τι εταιρικέ σχέσει δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και εργάζεται τώρα στο Ινστιτούτο Δημόσια Δίκηση τη Μαστρίχτη, όπου συμμερίζεται τη γνώμη του με του εργαζόμενους στον τομέα αυτό και έχει παρουσιαστεί ως εξπέρ της συνεδριάσεις μας στο παρελθόν. <clears throat> με μεγάλη χαρά λοιπόν για 10 λεπτά σου δίνω το λόγο. κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτέ. Στα αγγλικά θα μιλήσω, αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα στα γαλλικά προηγουμένω. Ο στόχος του Ιδρύματος για τη Δημόσια Δίκηση της Μαστρίχτης είναι η προώθηση της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης που θα περιλαμβάνει και καλύτερη κατανόηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και καλύτερη εφαρμογή τους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που, μας, που με καλέσατε για να λάβω το λόγο ενώπιον της Επιτροπής σας. Θα ξεκινήσω με μια, μια σειρά διαφανειών, αλλά δεν θα αναφερθώ στις διαφάνειες, γιατί είναι μακροσκελής. Θέλω να ξεκινήσω με το να θέσω μερικά θεμελιώδη ερωτήματα τα οποία πιστεύω ότι η Επιτροπή σας θα πρέπει να λάβει υπόψη και να απαντήσει. <clears throat> Δύο πράγματα καταρχήν. Τι δεν καλύπτει αυτή η οδηγία. Δεν αφορά την ελευθερία των δημοσίων αρχών για το πώς αποφασίζουν τη διεκχώρηση δημοσίων υπηρεσιών. Το πλήρες φάσμα από την άμεση παροχή υπηρεσιών μέχρι την απόλυτη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών είναι πάντα διαθέσιμο. Δεύτερον, η οδηγία αυτή δεν αφορά την οικονομική και πολιτική απόφαση του κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμόζονται δημόσια τέλη στην παροχή των ε, δημοσίων υπηρεσιών ή αν πρέπει να καλύπτονται μονάχα από τους φόρους. Η οδηγία αυτή εστιάζει την προσοχή της στο κατά πόσο η διάφανη και ανταγωνιστική διαδικασία εκχωρήσεων μπορεί να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο με τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται και δεύτερον το ερώτημα είναι κατά πόσον οι συμβάσεις εκχωρήσεων είναι διαφορετικές από τις υπόλοιπες δημόσιες συμβάσεις. Η νομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή δίνει την εντύπωση ότι είναι, γιατί είναι διαφορετικοί κανόνε που διέπουν αυτά τα δύο είδη συμβάσεων. Όλα αυτά προκύπτουν από την ιδέα ότι υπάρχει μια θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των συμβάσεων εκχωρήσεων και των άλλων συμβάσεων για προμήθεια αγαθών, παραδείγματο χάρη. Και αυτό μας οδηγεί σε δύο δευτερεύοντα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κάποια ανάγκη για την απονομή συμβάσεων εκχωρήσεων να ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν ναι, τι είδους ρύθμιση απαιτείται. Για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε κατά πόσο χρειάζεται παράγωγο δίκαιο για τα θέματα αυτά, <clears throat> υπάρχουν τρεις ε, σκέψεις που πρέπει να πριτανεύουμε. Καταρχήν, είναι ικανοποιητικό το πλαίσιο για την απονομή συμβάσεων εκχωρήσεων. Προς το παρόν, η Κομισιόν στην έκθεση αντικτύπου έδειξε ότι κατά την άποψή της αυτό δεν ισχύει ότι υπάρχει πολυμορφία εφαρμογή στα διάφορα κράτη-μέλη, υπάρχει ανεπαρκής νομική προστασία των διαγωνιζομένων, γιατί επειδή δεν καλύπτονται από την οδηγία οι εκχωρήσει για τις δημόσιες συμβάσεις, αυτοί που δεν είναι ικανοποιημένοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ε, αριστούν της οδηγία για τις νομικές θεραπείες και τέλος υπάρχει ανεπαρκής νομική κάλυψη γιατί το Ευρωπαϊκό <clears throat> Δικαστήριο σε διάφορες ε, υποθέσεις ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει σημαντικό τμήμα ενός περιορισμένου κινδύνου για να παρεμβεί ως δικαστήριο. Έχουμε επιπλέον το στόχο της Ευρώπης 2020, η οποία περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους επίτευξης της εσωτερικής αγοράς με την ανάπτυξη ενεργειακών δικτύων, δικτύων μεταφοράς και ψηφιακών δικτύων. Η ατζέντα της ε, σύνδεσης της Ευρώπης βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. <clears throat> Όπως τονίζει και η πρόταση της Κομισιόν, 60% αυτών των εταιρικών σχέσεων είναι ουσιαστικά στα πλαίσια των συμβάσεων εκχωρήσεως. Μιλάμε λοιπόν για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συμπλήρωση της ενιαίας αγοράς και για την Ευρώπη του 2020 και τα μεγάλα ποσά τα οποία συνδέονται με τα σχέδια της Ευρώπης 2020, η ατζέντα διασύνδεσης της Ευρώπης, 1,5 με 2 3 εκατομμύρια ευρώ θα γίνουν ακόμα πιο, πιο μεγάλα αυτά τα ποσά εάν δεν εξασφαλιστεί ότι διαλέγουμε την πιο αποδοτική σε σχέση με το κόστος λύση. <clears throat> Η Κομισιόν έχει τονίσει ότι οι εναλλακτικέ λύσεις θα ήταν με την ομολογία να επιλύονται προβλήματα τα οποία ανακύπτουν η Κομισιόν να ξεκινά διαδικασίες επί παραβάση να έχει μια νέα ανακοίνωση για την ερμηνεία της νομοθεσίας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν πολλά συμβόλαια υψηλής αξίας που δεν υπόκεινται στο παράγωγο δίκαιο μπορούν μονάχα να θεωρηθούν μη ικανοποιητικά από την άποψη αυτή από την Κομισιόν. Θα έπρεπε να θέσουμε το ερώτημα λοιπόν, τι είδου παραγωγό δίκαιο θέλουμε να έχουμε. θέλουμε να έχουμε μια πρότυπη οδηγία όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μήπως θα ήταν καλύτερο να ενσωματώσουμε και περαιτέρω κανόνες για τη συμβάση εκχωρήσεων στην τωρινή σύμβαση για τα στην τωρινή οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις. Φαίνεται ότι αυτή ήταν η άποψη που πριτάνευε στην, ε, το προηγούμενο φθινόπωρο. Και το τρίτο ερώτημα είναι μήπως τα συμβόλαια εκχώρησης θα πρέπει να υπόκειται στις ίδιες διαδικασίες απονομής όπως όλες οι υπόλοιπες δημόσιες συμβάσεις. Κάτι το οποίο η Κομισιόν δεν το απεδέχθη και το έχει αποκλείσει για τα συμβόλαια, για τις συμβάσεις ε, εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για να συνοψίσω η ιδέα του να έχουμε διαφορετικές διαδικασίες για τις εκχωρήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται αν θεωρήσετε ότι αυτού του είδους οι συμβάσεις εκχωρήσεων είναι πολύ διαφορετικές από τις άλλες δημόσιες συμβάσεις. Τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ομοιότηση. Είναι ε, συμβόλαια τα οποία οδηγούν σε μια κερδοφόρα σχέση. Έχουν επίσης μια αμοιβαία οικονομική σχέση οικονομικών φορέων. Πρέπει να εφαρμοστούν και συμβάσεις εκχωρήσεων βασικές αρχές για τις δημόσιες συμβάσεις και πρέπει να εξασφαλιστεί η καλύτερη σχέση απόδοσης κόστους. Επομένως υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Αν δει κανεί τώρα τα επιχειρήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί και στη διαβούλευση και αλλού. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να δικαιολογήσουν διαφορετικούς κανόνες για, τα, για τις συμβάσεις εκχωρήσεων, είχαν μεγάλη δυσκολία να επιχειρηματολογήσουν διαφορετικούς κανόνες γιατί είναι διαφορετική η ευθύνη του αυτού ο οποίος αναλαμβάνει την εκχώρηση. Αυτό μπορεί να δικαιολογεί διαφορετικούς όρους της συμβάσης αλλά όχι διαφορετική διαδικασία απονομής είναι το ποιος πληρώνει το φασιστικό. Όχι. Γιατί μπορείτε να, να έχετε εκχωρήσεις οι οποίες καλύπτονται από τους φορολογούμενους, από το Δημόσιο Ταμείο. Είναι ο τρόπος διαπραγμάτευσης διαφορετικός. Όχι, γιατί ο διάλογος, ο ανταγωνιστικός διάλογος δίνει τη δυνατότητα συζήτηση όλων των πτυχών των συμβάσεων με τους υποψήφιους. Και η διαδικασία διαπραγμάτευσης δίνει, η νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης του κανόνες για τις δημόσιε συμβάσει δίνει ακόμα περισσότερο. Παραβιάζεται με τους κανόνες αυτούς η επικουρικότητα. Όχι περισσότερο από ό,τι από άλλους ευρωπαϊκούς κανόνες και ιδίως για τους κανόνες για τις δημόσιε προμήθειε. Παραβιάζουν το πρωτόκολλο 26 για τι συνθήκε για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίζουν δηλαδή την ε, ε, ικανότητα των υποεθνικών ε, αρχών να οργανώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν όπως θέλουν. Όχι. Το μόνο πράγμα που κάνουν είναι ότι καθορίζουν τους κανόνες οι οποίοι ισχύουν όταν αποφασίσουν οι δημόσιες αρχές ότι μια εκχώρηση είναι η καταλληλότερη φόρμουλα που μπορεί να ακολουθηθεί. Τέλος, οι διάφοροι αυτοί κανόνες θα εμποδίσουν τη λειτουργία των εκχώρησεων. <clears throat> Αυτό είναι το κύριο θέμα υποσυζήτηση. Η διαδικασία διαβουλεύση το έκανε σαφές ότι περίπου 35 με 45% αυτών που απάντησαν στην έρευνά μας ξέραν ότι υπήρχαν άμεσες εκχωρήσεις. Και η Κομισιόν σε σχέση με την έρευνα για την νομική θεραπεία τόνισε ότι οι παράνομες απονομές ήταν ένα από τα κυριότερα προβλήματα τα οποία είχε να αντιμετωπίσει. Συνοψίζω λοιπόν. Το να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για, συμβόλαια, για συμβάσεις εκχωρήσεων είναι δύσκολο να το δικαιολογήσει κανείς. Και επειδή υπάρχουν πολλές ομοιότητες, το βάρος της απόδειξης είναι με τη μεριά αυτών που θέλουν να αποδείξουν ότι χρειάζονται χωριστοί κανόνες. Κατά τη δική μου άποψη, ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και να απαντήσει στα ερωτήματα της Κομισιόν είναι να υπόκεινται οι δημόσιες συμβάσεις εκχωρήσεων στις ίδιες διαδικασίες όπως και οι δημόσιες προμήθειες. Έχω κάποια ειδικά σχόλια για την οδηγία που ισχύει τώρα που μπορούμε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Έχουν να κάνουν με καλύτερη νομική προστασία και διαφάνεια, αλλά κατά την άποψή μας η συγχώνευση των ρόλων για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις εκχώρησης είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει δείξει η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπέρνατ για τις πολύ σαφείς σας ε, δηλώσεις. Επειδή αναφερθήκατε στην πρόταση της Επιτροπής, να καλωσορίσω την Τζοάννα Σικόφκα, η οποία είναι επικεφαλής της ομάδας της ε, Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και ελπίζω ότι θα παρεμβαίνετε κι εσείς αργότερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ξεκινήσατε την ακρόασή μας με τόσο σαφή και άμεσο τρόπο. Και τώρα να σας παρουσιάσω τον επόμενο μιλητή μα τον κύριο Πλάσμαν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπηρεσιών Γενικού Ενδιαφερόντος Κοινοφελών Υπηρεσιών και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εργοδοτών Επιχειρήσεων Κοινοφελών Υπηρεσιών. Για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να εστιάσω την ε, σύντομη παρέμβασή μου λέγοντας ότι εδώ και 13 χρόνια εργάζομαι μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα των συμβάσεων και θέλω να τονίσω τη σημασία της ε, ισοδικίας και της σωστής διαδικασίας στα πλαίσια αυτών των 13 χρόνων που παρατήρησα από την πλευρά της Κομισιόν. Το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να θίξω είναι η ανάγκη να υπάρξει μια οδηγία για τις εκχωρήσεις. Αν αναλύσει κανείς το κείμενο αυτό βρίσκει σαν συμπέρασμα ότι υπάρχει, ένας, υπάρχει ένα πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής που καλύπτεται από αυτή την οδηγία και αυτό το πεδίο εφαρμογής θα έπρεπε ήδη να έχει αντιμετωπιστεί με καλύτερο τρόπο από την έκθεση αντικτύπου. Πρέπει όμως να επενέσω και την Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν ανέλαβε αυτό το δύσκολο έργο που καλύπτει πάρα πολλού οικονομικού τομεί και πάρα πολλέ περιοχές εφαρμογή, προσπαθώντας να καταλήξουμε σε μια ευέλικτη διαδικασία, η οποία από τη μία πλευρά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα του θέματος, ε, και εκεί θέλω να εξάρω το έργο της Κομισιόν, ακόμα και αν έχω σε μεμονωμένα στοιχεία επικρίσεις, νομίζω το επέτυχε αυτό σε σημαντικό τρόπο, βαθμό θετικά μπορεί κανείς να επανέλθει σε θέματα χάρη για τα, τις τιμές κατοφλίων ή για την, ε, το μήκος της διαδικασίας παραχώρησης μιας σύμβασης, αλλά εμείς θα θέλαμε να υπάρξει και περισσότερη αντιμετώπιση ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων, ορισμένων εξαιρέσεων. Αλλά <clears throat> αυτές είναι εξαιρέσεις. Απλώς εν γέννη η Κομισιόν έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο είναι πολύ θετικό και με μικρές προσαρμογές θα μπορούμε να έχουμε μια πλήρη λύση για ένα ευρύτατο τομέα εφαρμογής. Για τις επικριτικές τώρα σκέψεις. Πρώτα απ' όλα είναι ιδιαίτερα ευρία η αντιμετώπιση της Κομισιόν και λείπουν δύο κριτήρια τα οποία ε, χαρακτηρίζουν τις συμβάσεις εκχωρήσεων. Καταρχήν, ότι η απονέμουσα αρχή παραμένει πάντα υπεύθυνη για την παροχή της υπηρεσίας που έχει εκχωρήσει σε κάποιον, ε, κάποια εταιρεία ή κάποιο άτομο. Και δεύτερον, ότι υπάρχουν πάντα αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία παίρνει αυτός ο οποίος αναδέχεται μία εκχώρηση του είδους αυτού. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι πολλές παροχές υπηρεσιών ε, θα μπορούσαν να είναι τμήματα συμβάσεων εκχωρήσεων και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι υπάρχουν παραδοσιακοί κανόνες και παραδόσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το ευρύ αυτό πεδίο εφαρμογής. Εμείς προσπαθήσαμε μαζί με την πόλη της ε, κολονίας να καταρτήσουμε ένα κατάλογο τομέων που μπορεί να καλυφθούν από αυτή την οδηγία. Καταλήξαμε στο γεγονός ότι παραγωγικά τα δίκτυα διανομής για ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, την εξαποστάσεως θέρμανση μπορεί να περιληφθούν, η υδροδότηση, η, ε, η υπόνομη, η αποκομιδή των σκυβάλων, οι λιμενικές και αεροπορικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, υγειονομικές υπηρεσίες, Ακόμα και πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες μπορούν να είναι αντικείμενο αυτών των ε, συμβάσεων εκχώρησης. Και κανείς φυσικά δεν είναι πλήρως έτοιμος για όλα αυτά τα θέματα. Για τις κοινωνικές υπηρεσίες εξάλλου η Κομισιόν έχει καταρτήσει, έχει προτείνει ένα κατάλογο πεδίου εφαρμογής, αλλά <clears throat> για αυτούς τους τομείς παροχής υπηρεσιών ισχύει και η οδηγία για τα ένδικα μέσα τα οποία μπορούν να τύχουν να, να τα επικαλεστούν αυτοί οι οποίοι είναι αναδοχοί εκχωρήσεων. Συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες έχουμε συζητήσει περισσότερο, είναι το θέμα των δικτύων διανομής, παραδείγματος χάρη δίκτυα στη Γερμανία και στη Γαλλία, όπου εδώ, στην περίπτωση αυτή, όταν γίνεται η εκχώρηση αυτή των δικτύων διανομής σε τρίτους φορείς, οι ενεργειακές <clears throat> εταιρείες χάνουν την άμεση επαφή με τους ε, πελάτες πια και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φανεί σαν σημαντικό πρόβλημα και στις δύο χώρες. Και εξάλλου ε, μπαίνουν νέοι παίκτες μεσαγωγικά στην αγορά, σε μια αγορά η οποία είναι εύθραστη πολλές φορές. Στη Γερμανία υπάρχουν πολλοί δήμοι οι οποίοι χάνουν έτσι την, ε, τον έλεγχό τους για τα δίκτυα διανομής και με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ασκήσουν πια ενεργειακή πολιτική σε επίπεδο Δήμου και κοινοτήτων, κάτι για το οποίο υπάρχει αίτηση από τους πολίτες. Επίσης για τις υπηρεσίες ευμάρειας, τις κοινωνικές παροχές, υπήρξε πρόσφατα μια έκθεση η οποία μια έρευνα που διενεργήθηκε στην Σουηδία, η οποία <clears throat> άνοιξε πολλές υπηρεσίες στον ανταγωνισμό και προχώρησε σε μια ανάλυση των αποτελεσμάτων και το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης είναι ότι υπήρξαν ελάχιστα μονάχα <clears throat> θετικά αποτελέσματα από, την, ε, από το άνοιγμα αυτών των υπηρεσιών στον ανταγωνισμό και επομένω υπάρχουν πολλές συζητήσει στη Σουηδία για το κατά πόσο είναι πρόσφορες αυτές οι υπηρεσίες για άνοιγμα στον ανταγωνισμό και όλα αυτά μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέροντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. <clears throat> για την υδροδότηση θα ακούσετε από τον συνάδελφό μου σε λίγο. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές θέσει σε διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ιταλία υπάρχει μεγάλη πίεση για το άνοιγμα στον ανταγωνισμό της υδροδότησης Άρα εκεί όμως έχουμε ειδικέ καταστάσεις. Ενώ στις ε, κεντρικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο βόρειες περιοχές όπως είναι η Αυστρία, η Γερμανία, οι κάτω χώρες δεν υπάρχει θέληση για άνοιγμα στο ανταγωνισμό της υδροδότησης και δεν είναι δημοφιλής μια τέτοια ιδέα γιατί θεωρείται το νερό σαν ένα δημόσιο αγαθό το οποίο δεν πρέπει να υπόκειται στον ανταγωνισμό. Υπάρχουν και περαιτέρω στοιχεία τα οποία μπορούν να δώσουν λαδί σε επικρίσει. Δεν πρόκειται να τα διεξέλθω όλα. Θα σταθώ μόνο σε ορισμένα. Πρώτα απ' όλα, μέσω τη οδηγία αυτή, πολλοί τομεί ανοίγονται στον ανταγωνισμό, χωρίς όμως προηγουμένως να υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο, το νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτοί οι τομείς. Αυτό οδηγεί, όπως είδαμε στην περίπτωση της αποκομιδής των σκουπιδιών σε πολλές διαμάχες και προβλήματα. Και ιδίως στον τομέα της ενέργειας είδαμε να προκύπτουν αρνητικά αποτελέσματα το να υπάρχει μια αγορά με πολλούς εμπλεκόμενους, πολλούς παίκτες <clears throat> και να υπάρχουν νέοι παίκτες οι οποίοι θα μπουν σε μια νέα αγορά πολλές φορές οδηγεί σε ασάφεια και σύγχυση. Το βασικό στοιχείο αυτής της οδηγίας, <clears throat> κατά την άποψή μου, είναι το ότι η Κομισιόν προτείνει να υπάρξει και η εφαρμογή της οδηγίας για την, ε, τα 11 μέσα ή καλύτερα τις νομικές θεραπείες στην περίπτωση των εκχωρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν οι, οι, τρίτε, τρίτοι φορείς να κάνουν ε, προσφυγές για τα θέματα αυτά και στη Γερμανία υπάρχει μεγάλη πίεση στα δικαστήρια από τις προσφυγές αυτές και αυτό δεν ε, βοηθά την αποτελεσματικότητα της απόδοσης της δικαιοσύνης. Και τίθεται εδώ και σε ε, ένα αμφιβόλο και η δυνατότητα των πολιτικών να αποφασίζουν και όχι των δικαστηρίων στη θέση τους. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο ορισμό του τι είναι οι συμβάσεις εκχωρήσεων και επίσης να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στις ενδεχόμενες εξαιρέσεις. Παραδείγματο χάρη, όλος ο τομέας του, της υδροδότησης να παραμείνει εκτός των συμβάσεων αυτών εκχωρήσεων. Δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή αγορά ύδατος, ενιαία αγορά, ούτε υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί μια αγορά εκχωρήσεων. Οι κοινωνικές ε, υπηρεσίες, οι υγειονομικέ, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να παραμείνουν έξω από αυτή την οδηγία. Και επίση οι υπηρεσίες αστικών μεταφορών ο κανονισμός 1370 του 2007 θα πρέπει να παραμείνει αυτός ο οποίος διέπει τις ε, συγκοινωνίες αυτές. Κάποιες ακόμα συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες όμως δεν θα τις αναφέρω τώρα. Μπορείτε να τα δείτε βέβαια στη διαφάνειά μου αν θέλετε. Απλώς θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο ακόμα που είναι η έννοια των υπηρεσιών in-house που παρέχονται από τον ίδιο το φορέα. Εδώ έχει παρουσιάσει πολύ καλές προτάσεις η Κομισιό. Και υπάρχει το θέμα του δευτέρου, του δεύτερου, του δεύτερου χαρακτηριστικού, του δεύτερου τέκελ όπως λέγεται, που λέει ότι 90% των υπηρεσίων θα πρέπει να παρέχονται στους, ε, στις υπηρεσίες μάλλον στον χώρο ο οποίος είναι υπό τον έλεγχο των δημοσίων αρχών θα ήταν η σωστή διατύπωση. Και θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής, ότι η Κομισιό μας έχει πει πάντα στο παρελθόν και το έχουμε πιστέψει μέχρι στιγμής, <clears throat> ότι αυτή η οδηγία για την παροχή υπηρεσιών, για, την, για τις εκχωρήσεις, θα έπρεπε να έχει το στόχο σε περιπτώσεις που υπάρχει προσπάθεια εξωτερήκευσης και outsourcing για τις ε, υπηρεσίες αυτές να καλύπτονται από μια οδηγία. Αν πράγματι αυτός είναι ο κύριος στόχος αυτής της ε, διαδικασίας και μπορεί να περιλαμβάνει και τις εξωτερικευμένες υπηρεσίες και την, ε, τις υπηρεσίες in-house, τότε μπορούμε ίσως να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Μία μήνα στα 10 λεπτά μου. Είμαστε γενναιόδοροι, διότι καθυστερήσαμε τον προηγούμενο μιλητή λίγο. Λοιπόν, επόμενη ειδικό ε, για τις εκχωρήσεις, η Μπριγκίτα Σιμών, από την Βίνση. Για 10 λεπτά έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτή την ακρόαση. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για τη δραστηριότητα εκχώρηση του δικού μα ομίλου. Στην παρουσίασή μου θέλω να επικεντρωθώ σε μερικά σημαντικά σημεία, γιατί δεν μπορώ να καλύψω προφανώ όλα τα θέματα που, ναι, που εγείρει αυτή η πρόταση οδηγία. Ήθελα λοιπόν εδώ να σταθώ στον ειδικό χαρακτήρα των εκχωρήσεων. Κάτι που ήθελε να καλύψει αυτή η οδηγία. Δυστυχώ η πρόταση οδηγία δεν ανταποκρίνεται στον προαναγγελθέντα στόχο. Και αυτό για του εξή λόγου. Πρώτα απ' όλα, ούτε στην ουσία ούτε στη μορφή της δεν ε, αποτελεί μια ήπια προσέγγιση. Έπειτα αφορά την απονομή των εκχωρήσεων αλλά και την εκτέλεση καθώς και το καθεστώς προσαρμογής τους και θα επανέλθω σε αυτό και ουσιαστικά πρόκειται για ένα copy-paste της πρότασης οδηγίας για τους δημόσιους διαγωνισμούς αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση. Θα ήθελα να σταθώ σε τέσσερα βασικά σημεία. Το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, του ορισμού τη αξία και τη διάρκεια τη εκχώρηση, που είναι σημαντικέ έννοιε, την διαδικασία απονομής και τέλο το καθεστώ προσαρμογή ή μετατροπή. Για το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία υπάρχει προφανώ μια σοβαρή αντίφαση μεταξύ του στόχου που προαναγγέλλεται για, ε, για του διαγωνισμού εκχωρήσεων και των όρο που προβλέπονται τελικά. Στα, άρθρα 11 και 15 μιλάμε για τομεί δραστηριότητε που έχουν να ε, κάνουν με, τους, με τις εκχωρήσεις και οι οποίες αντιμετωπίζονται ανταγωνιστικά. με πολλές βέβαια εξαιρέσεις. Το άρθρο 11 αναφέρεται στην, ε, σε διάταξη της οδηγίας για τους ειδικούς τομείς και σε τομείς ε, κοινών υπηρεσιών με ειδικά ή εξαιρετικά δικαιώματα. Αυτό επιτρέπει στους κρατικούς φορείς να αναθέσουν ε, σοβαρές αρμοδιότητες χωρίς όμως να υπάρχει χωρίς να υπάρχει ανταγωνιστικότητα περιορισμός διάρκειας στους φορείς που συνδέονται με διάφορες εταιρείε. Το άρθρο 15 μιλάμε για τις υπηρεσίες in-house με εξαιρέσεις, εξαιρέσεις που τις επιτρέπει και η νομολογία. Με το άρθρο αυτό οι δημόσιοι φορείς μπορεί να θεωρήσουν απλούστερο να, να τρέξουν σε έναν φορέα in-house και να μην διοργανώσουν διαδικασία για μια, ένα διαγωνισμό. Αυτό έχει να κάνει και με την δικαστική απόφαση Κακάλ. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ λίγο στην αξία και τη διάρκεια των εκχωρήσεων, κάτι που είναι σημαντικό. Η αξία που επαναλαμβάνει η διάταξη των δημοσίων διαγωνισμών εξαρτάται από υπολογισμού για τα έργα και τι υπηρεσίε, αλλά δεν διευκρινίζεται ο τρόπο που θα γίνεται η διάκριση μεταξύ των εκχωρήσεων έργων και εκχωρήσεων υπηρεσιών. Η διάκριση όμω αυτή μπορεί να είναι πηγή δυσκολιών για του δημόσιου φορεί στο βαθμό όπου οι εκχωρήσει έργων πάντοτε συνοδεύονται από υπηρεσίε και αντιστοίχω ε, οι εκχωρήσει υπηρεσιών συνοδεύονται από έργα. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να εφαρμόζεται ένα απλό κανόνα και για τις δύο περιπτώσεις, ε, έργα και υπηρεσίες. Να βασιζόμαστε στον κύκλο εργασιών και την υπολογιζόμενη διάρκεια της εκχώρησης. Ως προς την διάρκεια της εκχώρησης, αυτή δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη είναι τα ποικίλα χαρακτηριστικά μιας εκχώρηση. Όπως έχει λοιπόν ε, διατυπωθεί ο ορισμό μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στι εκχώρησει έργων, με την έννοια της επένδυσης. Όμως η διάρκεια μιας σύμβασης εκχώρηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την επίτευξη των στόχων, τι ε, ε, τις επιδόσεις μάλλον, την ποιότητα που όλα αυτά υλοποιούνται σε μια διάρκεια χρόνου. Επίση, υπάρχει πρόβλημα με τη σημερινή διατύπωση, διότι καλύπτονται μόνο οι επενδύσει που γίνονται κατά τη στιγμή τη εκμετάλλευση, τη πραγματοποίηση ε, των έργων ή τη ε, παροχή των υπηρεσιών και όχι των ε, υπόλοιπων διαδικασιών και δραστηριοτήτων που μπορεί να αναλάβει ο υπεύθυνο της εκχώρηση. Για την απονομή τώρα, θα ήθελα να σταθώ στα εξή σημεία. Τι διαπραγματεύσει, τι τεχνικέ διευκρινήσει και τη διαδικασία απονομή την ίδια. Για τι ε, διαπραγματεύσει που θα διοργανώνονται. Εδώ χαιρετίζω την επιλογή που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να δίνεται προτεραιότητα στι διαπραγματεύσει στο πλαίσιο των αναγκών διαφάνεια και χνηλεσιμότητα παρά να απονέμονται με ανταγωνιστικό διάλογο οι διάφορες εκχωρήσεις. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να είναι πολύ σαφέστερη η επιλογή των, ε, της εκχώρησης και δεν θα πρέπει η διαδικασία αυτή απονομής να θεωρείται αναγκαία. Διότι ο όρο αναγκαία και μόνον δίνει δικαίωμα για πολλέ ερμηνείε. Τώρα για τις ε, τεχνικέ διευκρινήσει, το κείμενο αυτό ακριβώ έχει αντιγραφεί από το σχέδιο κειμένου για του δημοσίου διαγωνισμού. Εκεί όμω έχουμε να κάνουμε και με φορεί τοπική αυτοδιοίκηση. κάτι που δεν ισχύει εδώ. Ε, δεν μπορεί να επιβληθούν τα ίδια μέτρα στις εκχωρήσεις ε, στο σύνολό τους, διότι εδώ το στοιχείο του κινδύνου το αναλαμβάνει ο υπεύθυνο τη εκχώρηση. Αυτό είναι κεντρικό στοιχείο του ορισμού. Οι εκχωρούντε λοιπόν ε, πρέπει να ανταποκριθούν στι ανάγκε που επιβάλλονται από τι δικέ του τεχνικέ επιλογέ και να απολογηθούν στο δημόσιο φορέα ή του φορεί τοπική αυτοδιοίκηση, εφόσον χρειαστεί, να λογοδοτήσουν δηλαδή. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει στάθμιση των κριτηρίων ή ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Αυτές οι μέθοδοι όμως δεν μπορεί να αρμόζουν ε, στις εκχωρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή. Τώρα σε ένα επίσης σοβαρό θέμα το καθεστώς ε, μετατροπής ή προσαρμογής των εκχωρήσεων. Όπως το έλεγα, η οδηγία στον τίτλο της αναγγέλει μια, διαδικασία, μια οδηγία περί της διαδικασίας απονομής αλλά τελικά καλύπτει και το καθεστώ εκτέλεση. Μια πρώτη διαπίστωση για την ουσία, για το θέμα τη μετατροπή ή προσαρμογή, είναι ότι το κείμενο είναι τελείω ανάρμοστο σε σχέση με τι ανάγκε των εκχωρήσεων και δεν καλύπτει τι επιτακτικέ ακριβώ Είναι ανάρμοστο για το καθεστώς ε, των εκχωρήσεων και τη μεταβλητότητα της σύμβασης, τη μεταβλητότητα των υπηρεσιών δεν την καλύπτει η σημερινή διατύπωση. Αυτά είναι υποκείμενα της έννοιας της σύμβασης της ίδιας για τις εκχωρήσεις. Εδώ έχουμε αντιγράψει το κείμενο του άρθρου 42 του σχεδίου το άρθρο μάλλον 72 από το σχέδιο κειμένου για του δημόσιου διαγωνισμού, ε, Είναι πανομοιότυπο με το άρθρο 44 του οδηγίας που κοιτάζουμε και βεβαίω έχει να κάνει και με την ομολογία του ΔΕΚ. Όμω, ε, τα πράγματα εδώ με τι εκχωρήσει είναι διαφορετικά σε σχέση με του δημόσιου διαγωνισμού, τι δημόσιε συμβάσει, ιδίω ω προ την εκτέλεση. Διότι στι ε, δημόσιε συμβάσει μιλάμε για μακροπρόθεσμε εταιρικέ σχέσει με διάρκεια που μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν πρόκειται για, ε, την, ε, για κατασκευαστικέ συμβάσει, όπω αυτοκινητοδρόμων. Εκεί αρχικά χρειάζεται ευελιξία στις εκχωρήσεις, διότι θα πρέπει στη διάρκεια να μπορεί να μετατραπεί η σύμβαση, να προσαρμοστεί στις ρυθμιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Θα μπορούσα να δώσω το παράδειγμα ως προς τη ρυθμιστική εξέλιξη την οδηγία για την ασφάλεια των σειράγων που έχει να κάνει με την ασφάλεια των αυτοκινητοδρόμων. Κάτι που μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, αλλά αφορά και σοβαρά ποσά. Είναι λοιπόν σημαντικό οι συμβάσεις εκχωρήσεων μεγάλης διάρκειας να μπορέσουν να αναπνεύσουν, γιατί μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες μέχρι να ολοκληρωθούν, ιδίω τι εκχωρήσεις ε, έργων που μπορεί να είναι πολύ μεγάλη πραγματικά η χρονική διάρκεια και επίσης πολύ σοβαρές οι επενδύσεις που εμπλέκονται. Ως προς την μορφή τώρα, το άρθρο αυτό όπως το έχουμε στα χέρια μας είναι τελείως ανέφικτο να εφαρμοστεί, διότι όπως έλεγα και προηγουμένως, το άρθρο αυτό έχει αντιγραφεί τελείως από την, ολόκληρο από την ε, οδηγία για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Ε, οι όροι ε, των δημόσιων συμβάσεων δεν μπορεί να ισχύουν και για τις εκχωρήσεις. Το κείμενο ανατρέχει διαρκώς τον όρο τιμή. Τιμή της σύμβαση, τιμή της εκχώρησης. Όμως στις εκχωρήσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Θα έλεγα πολύ απλά να αλλάξουμε τον όρο με τον όρο αξία. Κάτι που έχει να κάνει και με τον ορισμό της αξίας που αναφέραμε προηγουμένως υπό το άρθρο 6. Προτείνουμε λοιπόν να αντικατασταθεί απλώς στο κείμενο ο όρος τιμή με τον όρο αξία και θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακριβώς στην αξία το όριο του 50% που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου ως προς την μετατροπή. Σε ό,τι αφορά τις εκχωρήσεις έργων που όπως έλεγα προηγουμένως θα πρέπει να διακρίνονται από τις εκχωρήσεις υπηρεσιών δεδομένου της μεγάλης τους διάρκειας, του ποσού των επενδύσεων που μπορεί να απαιτούνται. Θα έλεγα ότι πρέπει να ισχύει αυτό το ανώτατο όριο του 50% για το συνολικό ποσό της εκχώρησης, ανάλογα όμως με τις ημερομηνίες μετατροπής που ε, μπορεί να προβλέπονται. Για να ολοκληρώσω, θα έλεγα ότι το κείμενο που εξετάζουμε είναι, παρουσιάζει ένα πραγματικό κίνδυνο προς την εσωτερική αγορά, αντιφάσκει με τον αρχικά αναγγελθέντα στόχο και πρέπει να βελτιωθεί. Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των ε, συμβάσεων εκχωρήσεων που δικαιολογούν την ύπαρξη αυτή τη οδηγία, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει επαναστόχευση ω προ τον αρχικό σκοπό, δηλαδή την διαδικασία απονομή και να βεβαιωθούμε για την νομική ασφάλεια και το άνοιγμα τη αγορά των εκχωρήσεων στο επίπεδο τη Ένωση. Με συγχωρείτε που ήμουν τόσο ε, ταχύτητα, στην παρουσίασή μου, αλλά έπρεπε να μείνω στα 10 λεπτά. Well, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιμών, ευχαριστώ και του τρει ομιλητέ για τις παρουσιάσεις τους. Αν και δεν ήταν ταυτόσιμες. Αλλά αυτό είναι ακριβώς είναι το θέμα. Λοιπόν, τώρα οι ερωταπαντήσεις. Ο κύριος Γιουβέν πρώτος, Κοφεράτη, για να δω ποιοι είναι, Βαγέαν, Σκιώδης πρώτο Παντζέρη, Ρούλα, Μπουζόη άμετα στο δεύτερο γύρο. Τέλο να αρχίσουμε με τον κύριο Ζουβέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και του τρει ομιλητέ. Παρατηρώ ότι και οι τρει βασικά είναι υπέρ ενό ενοποιημένου συστήματος, διαφορετικού για τον καθένα. Η κυρία Σιμών κατέληξε λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνο να κλείσει η αγορά, ενώ ο κύριος Πασμάνη είπε ότι υπάρχει ο αντίθετος κίνδυνος υπερβολικού ανοίγματο. Να μην πέσουν όλα στο στίβο του ανταγωνισμού, είπε. Κύριε Μπάρνετ, κύριε Πλάσμαν, δεν πιστεύετε ότι αφού μιλήσατε για το νερό και τα λοιπά, δεν πιστεύετε ότι πέρα από οποιοδήποτε θεωρητικό, θεωρητικό ολική εξέταση του πράγματος, η ολική πολλές φορές απουσία κάθε συμβολέου, δεν μιλάω καν για ανταγωνισμό, αλλά οποιασδήποτε χώρηση είναι προβληματική. Εμείς στη Γαλλία ξέρουμε ότι υπήρξαν τεράστιες περιπτώσεις διαφθοράς και δωροδοκίας και γι' αυτό συζητήσαμε θέματα όρων της διαφάνειας. Αν συνεχίσουμε έτσι και λέμε ότι μπορούμε να δεχτούμε και την απουσία συμβολέων, νομίζω ότι θα συνεχιστεί το πρόβλημα. Ίσως οι εκχωρήσεις να πρέπει να ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τις δημόσιες προμήθειες, δεν ξέρω. Βασικό στοιχείο πάντως είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει αυτός που παίρνει το συμβόλαιο. Στο λοιπόν η κυρία Ρούλα και μετά άλλη σκιώδης. Θέλατε κι εσείς να μιλήσετε κύριε Παντσέρη τώρα ή μετά. Α, μετά ας πουμε Α, καλά το. Η κυρία Ρούλα λοιπόν. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι συντάκτρια γνωμοδότηση για την Περιφερειακή Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ήταν παρόντες σε αυτή την ε, πρώτη δημόσια ακρόαση για το θέμα αυτό, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία τέτοια ακρόαση και θέλω ιδίω να τονίσω ότι τρεις πρώτες ε, ομιλίες έδειξαν ότι είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο αυτό το σχέδιο οδηγίες. Και το ερώτημα μου είναι τι προσθέτει Τη υπομορφή αξία, τι δίνει στους πολίτες αυτή η πρόταση. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα πεπισμένη από αυτά τα οποία άκουσα. Δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου αυτή η πρόταση. Όλα ξεκινούν με τους ορισμούς. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, ομιλητέ να μου αναφέρουν πώς βλέπουν αυτοί το θέμα του ορισμού, τι είναι εκχώρηση, το θέμα τη ευθύνη, των αποκλειστικών δικαιωμάτων, της ανάληψης κινδύνου. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα που συνδέονται με τον ε, ορισμό. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι το θέμα του πεδίου εφαρμογής. Όταν μιλήσω σε σχέση με το θέμα αυτό και εδώ όλη την ε, πρόταση δεν παραμένει τίποτα το οποίο δεν καλύπτεται από την οδηγία. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς ακριβώς καθορίζεται το, το πεδίο εφαρμογής γιατί νομίζω ότι είναι υπερβολικά ευρύ όπως φαίνεται μέχρι στιγμής. Κυρία Φερχέιεν. Ευχαριστώ και εγώ να θέσω ένα ερώτημα και στους τρεις ομιλητές. Για μένα ένα από τα κύρια σημεία στην ε, παρέμβασή σας είναι το θέμα της διαφάνειας. Η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου πρέπει να εξασφαλιστεί με αυτή την οδηγία. Τώρα, λόγω των διαφορετικών αποφάσεων που υπάρχουν και των διαφορετικών μορφών συμβάσεων, μήπως θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Κομισιόν το γεγονός ότι υπάρχουν αποκλίνουσες ερμηνείες αυτού του δικαίου και αυτό δεν οδηγεί σε ασφάλεια δικαίου και δεύτερον μήπως οδηγούμε σε κάτι όπου το παράγωγο δίκαιο θα υπερ, υπερτερεί δηλαδή, του πρωτογενούς δικαίου. Παραβιάζεται λοιπόν η δυνατότητα κυριαρχίας των ε, αρχών σε διάφορους τομείς. Η ομιλήτρια είναι πολύ μακριά από το μικρόφωνο και θα πρέπει εδώ να υπάρξει και σεβασμός των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών ή των υποεθνικών αρχών να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Και για τον κύριο Μπερνέτ ιδιαίτερα πιστεύετε ότι με αυτή την οδηγία δημιουργείται περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη ασφάλεια δικαίου και αυτές οι διαδικασίες θα κάνουν πιο εύκολες τις εταιρικέ σχέσεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα ή θα τις κάνουν πολύ πιο δύσκολες για διάφορους δήμους και κοινότητες. Μια πιο βαριά διαδικασία χάρη για την προκήρυξη διαγωνισμών και οποιαδήποτε αλλαγή της ε, μια συμβάσεως θα πρέπει να περάσει πάλι από την επαχθή αυτή διαδικασία η οποία αναφέρεται στην οδηγία. Ποιες είναι λοιπόν οι συγκεκριμένες επιπτώσεις που θεωρείτε ότι θα υπάρξουν στις εταιρικές σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. και μήπω θα οδηγήσουν τελικά στου Δήμου και τι κοινότητε να μην κάνουν καθόλου συμβάσει εκχωρήσεων και να κρατάνε στα χέρια του όλε τι υπηρεσίε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κύριο Κομφεράτη. Ευχαριστώ. Νομίζω Ορθώς προσπαθεί η Επιτροπή να καθορίσει τις προϋποθέσεις ανάθεσης συμβάσεων εκχώρησης στην Ευρώπη. Όμως, η προσπάθεια της Επιτροπής έχει μερικές πιθανότητες να φτάσει στην επίτευξη του στόχου, αλλά πρέπει προηγουμένως να τεθεί σωστά το πεδίο εφαρμογή, να καθορίσουμε ποιε είναι οι εκχωρήσει. Οι εκχωρήσει είναι αυτέ που αναφέρονται μεν, αλλά με κάποιε προσθήκε. Το σύστημα εντροδότηση λόγου χάρη είναι δημόσιο ε, στις, και κρατικό στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορεί λοιπόν να περιλαμβάνεται στις εκχωρήσει. δεν μπορεί να προσφέρεται μια τέτοια υπηρεσία στους πολίτες με τις ίδιε προποθέσει. Αυτό ισχύει και κάποια άλλα δίκτυα όπως την ηλεκτρική ενέργεια. Ένα θέμα είναι η παραγωγή που μπορεί να υπόκειται σε οποιοδήποτε παρέμβαση ρυθμιστική, αλλά άλλο είναι η διανομή της. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας όπως την παραγωγή τη, τότε η εκχώρηση ουσιαστικά εδογεί σε ιδιωτικοποίηση που αποκλεί μέρο μέρος των πολιτών. Αυτές είναι προϋποθέσεις ώστε να μην γίνει η χρήση των εκχωρήσεων αυτών ανταγωνιστική στο όλο σύστημα, οπότε να μην υπάρξουν και τα πετούμενα έσοδα από τις εκχωρήσεις. Πρέπει λοιπόν η συζήτηση να περάσει σε ένα νέο ε, θέμα, δηλαδή τα όρια των ορισμών, το πλαίσιο που θέλουμε να καθορίσουμε και όχι μόνο το εσωτερικό αυτού του πλαισίου. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτές οι δημόσιε χωρίσει μπορεί να αλλάξουν ε, την ζωή εκατομμυρίων πολιτών. Είναι ένα θέμα ύψης της που πρέπει να απασχολήσει και τα θεσμικά όργανα και βεβαίω απασχολεί και του τελικού χρήστε. Well, uh, Ευχαριστούμε. ως σκιώδης εισηγητής για την έκθεση του κυρίου Ζουβά και ως πρόεδρος θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στην κυρία Μπερνέτ, στην πρώτη ομιλία που ακούσαμε. Στον κύριο Μπερνέτ, συγγνώμη. Ο κύριος Μπέρνετ είπε ότι η πρόταση που εξετάζουμε σκοπό έχει να ρυθμίσει και να διοργανώσει την εκχώρηση συγκεκριμένων συμβάσεων στο δημόσιο τομέα. Όχι όμω να ορίσει τι ακριβώ πρέπει να ρυθμιστεί. Αυτή είναι μια απόφαση που οι πελάτε στην ουσία θα πρέπει να λάβουν. Συμφωνώ, διαφωνώ λοιπόν ε, τελείω με τον κύριο Κομφεράτη που δεν με ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά θα το πω έτσι κι αλλιώ. Το σύστημα εντροδότηση στη χώρα μου είναι ιδιωτικοποιημένο. Και κύριε Κομφεράτη, δεν μπορεί η νομοθεσία να αποφασίζει τι είδου υπηρεσίε θα παρέχονται και τι όχι. Ε, διαφωνώ λοιπόν απολύτω μαζί σα και συμφωνώ με τον κύριο Κλάσμαν ότι αποστολή αυτού του κανονισμού θα πρέπει να είναι και τι θα περιλαμβάνεται. Θα έπρεπε να υπάρχει το νομικό πλαίσιο σε ένα πνεύμα ανταγωνιστικότητα. Η κυρία Σιμών είπε ότι δεν θα υπάρξει ανταγωνισμό με αυτή την πρόταση οδηγία. Μα δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο με τον εν κανονισμό. Πάντω θα δώσω σε όλους τους ομιλητέ μα δύο λεπτά ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν σε όσα άκουσαν και θα ξεκινήσουμε αντίστροφα με την κυρία Σιμών, μετά με τον κύριο Πλάσμαν και μετά με τον κύριο Μπέρνετ. Κυρία Σιμών, θέλετε να απαντήσετε πρώτη. Πάρα πολύ σύντομα, σε δύο λεπτά για το ερώτημα σε σχέση με τη νομική, με τη νομική ασφάλεια και τη διαφάνεια που προσφέρει το κείμενο. Αυτό ήταν και ο στόχο του, να εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια. Ξέρουμε ότι σε πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει σήμερα νομοθεσία η οποία να διέπει τι εκχωρήσει. Στη Γαλλία έχουμε εδώ και πολύ καιρό, όπω υπενθύμησε ο κύριο Ζουβέν, με το νόμο Σαπέν, μια ρύθμιση, αλλά υπάρχουν χώρες όπου ελείπει μια τέτοια νομοθεσία και ιδίως για την ε, εκχώρηση υπηρεσιών. Αλλά με το κείμενο έχει σήμερα, με τις πολλές ατέλειες που έχει σε επίπεδο διατύπωσης και σύνταξης, που οφείλονται στο γεγονός ότι μεταφέρονται διατάξεις που διαπούν τις αγορές στην περίπτωση των εκχωρήσεων, φοβάμαι πολύ ότι ο στόχος της ασφάλειας δικαίου δεν επιτυγχάνεται, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να προκύψουν ερμηνείες οι οποίες θα είναι αποκλίνουσες και αυτό δεν είναι και ο στόχος της οδηγίας. Πιστεύω το κείμενο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, οπότε πρέπει να γίνει ακόμα μια περαιτέρω επεξεργασία στο κείμενο για να επιτευχθεί αυτό και σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της αγοράς. Επιμένω ότι εμείς βλέπουμε κυρίως τον κίνδυνο να κλείσει αυτή η αγορά, διότι με, όλους αυτούς, με όλες τις ρήτες αποκλεισμού που περιέχονται στο κείμενο, υπάρχει πραγματικά ο κίνδυνος σε ένα μεγάλο μέρος δραστηριότητας να βρεθούν εκτός ανταγωνισμού και λόγω του κατοφλίου ε, του 90% που περιλαμβάνεται μπορεί η, αγορά να ξεφύγει τελείως από τον ανταγωνισμό, κάτι το οποίο δεν φαίνεται λογικό. Ο κύριος Πλάσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το ερώτημα του κυρίου Ζουβέν. Ε, για το αν μπορεί να υπάρξει απουσία προβλημάτων. Εγώ θα έλεγα ναι, όταν υπάρχει εξωτερήκευση σε ορισμένους τομείς, ε, αλλά κινδυνεύουν πάντα να υπάρξουν ε, προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν. Σε χώρες όπου υπάρχουν πολύ ισχυρέ τοπικές αρχές, η εκτέλεση εργασιών, η παροχή υπηρεσιών από από εξωτερικούς φορείς, αυτό φαίνεται σαν μια εκτέλεση υπηρεσιών υπό την αιγίδα του Δήμου. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό. Δεν είναι ακριβώς η περίπτωση της εξωτερήκευσης υπηρεσιών. Και για το ερώτημα της κυρίας Ρίουλε σε σχέση με τους ορισμούς, εγώ έχω δώσει την απάντησή μας. Εμείς θέλουμε να εμπλουτίσουμε αυτό τον ορισμό, δίνοντας το στοιχείο αυτό ότι η υπολοιπόμενη ευθύνη παραμένει στα χέρια του τοπικού φορέα, του Δήμου ή της κοινότητας και επίσης τονίζοντας ότι μια εκχώρηση δεν ε, σημαίνει πάντα αποκλειστικά δικαιώματα. Τώρα υπάρχει διαφορετική ε, εμπειρία σε άλλες χώρες, στο Λονδίνο παραγωγικα με τον υπόγειο σιδηρόδρομο που βλέπουμε ότι η ευθύνη για τον τομέα αυτό δεν είναι αυτού που ε, που ασκεί τι υπηρεσίε που λειτουργεί, παραδείγματο χάρη τον υπόγειο σιδηρόδρομο, αλλά παραμένει στα χέρια του, του Δήμου. Για τι δυσκολίε σε σχέση με την ασφάλεια δικαίου στην εφαρμογή αυτή τη οδηγία, θέλω να πω ότι επειδή είναι ευρύ το πεδίο εφαρμογή μαζί με του οδηγού, με του ορισμού που δίνονται και το γεγονό ότι σε πολλού τομεί υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν ακόμα επιδηθεί, όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Ευχαριστώ. Δεν απαντήσατε το δικό μου ερώτημα, κύριε Πλάσμαν, για την φιλοσοφία που διατρέχει αυτό το κείμενο. Εγώ είπα ότι ο αποκλεισμό ορισμένων τομέων εναπόκειται στην αρχή η οποία απονέμει τη συμβάση εκχωρήσεων και όχι στην νομοθεσία. είπατε στην παρουσίασή σας, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος, ότι θέλετε να προσθέσετε εξαιρέσεις στις συμβάσεις, ενώ η νομοθεσία πιστεύω ότι είναι για τη διαχείριση συμβάσεων και ότι είναι σίγουρα η ευθύνη των πελατών, των αρχών που απονέμουν, το αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν συμβάσει χωρίσεως και όχι να αναφέρεται στην ε, οδηγία. Ναι, ναι, ναι, εγώ διαφωνώ με τον κύριο Μπερνέτ. Νομίζω ότι έχετε απαντήσει εσείς ο ίδιος. ο κύριος Μπερνέτ. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα αυτά τα οποία πηγαίνουν προς τον πυρήνα της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει θέσει το βασικό ερώτημα για την οδηγία αυτή. Όχι ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να την χάνουν ρύθμισης, ούτε για την ελευθερία των τοπικών αρχών ή οποιοδήποτε δημόσιο φορέα να οργανώσει υπηρεσίες με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε όταν και εάν ληφθεί η απόφαση να προχωρήσουμε σε μια εκχώρηση. Και αυτό το τόνισε πολύ σαφώς η κυρία Σικόφσκα όταν μίλησε ενώπιον της Επιτροπής σας στις 6 Φεβρουαρίου από την πλευρά της Κομισιόν. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σαφές και βρισκόμαστε κοινότητα στον κύριο Σικόφσκα για τα συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν αυτό που είπε καταρχήν ο κ. Ναι, είναι δυνατόν να επιχειρηματολογήσει κανείς ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων εκχωρήσεων. Το ερώτημα είναι αυτό δικαιολογεί διαφορετικές διαδικασίες απονομής. Κατά τη δική μου άποψη υπάρχει διαφορετικός κίνδυνος στις δύο περιπτώσεις που δικαιολογεί διαφορετικούς όρους στη σύμβαση αλλά όχι διαφορετικές διαδικασίες απονομής δύο μονάχα εξαιρέσει που θα μπορούσατε να σκεφτείτε. Πρώτον, επειδή οι συμβάσεις εκχωρήσεων είναι μακρύτερε στο χρόνο από ότι οι δημόσιε συμβάσει θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο εύκολη διαδικασία τροποποίηση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στην περίπτωση μια εκχώρηση, ιδίω ακολουθώντα την αρχή που προέρχεται από, τον γαλλικό, από το γαλλικό διοικητικό δίκαιο της επανεξεσορρόπησης μιας σύμβασης όταν συμβούν γεγονότα ανωτέρας βίας. Επίσης για τα θέματα των κατοφλίων. Μπορεί κανείς να συζητήσει αν τα κατόφλια για τις ε, εκχωρήσεις θα πρέπει να είναι διαφορετικά από ό,τι για τις δημόσιες συμβάσεις. Για το θέμα που έθεσε η κυρία Γουίλα και η κυρία Φερχάιεν σε σχέση με την ασφάλεια δικαίου, όταν έκανα μια λεπτομεριακή ανάλυση αυτής της οδηγίας, κατέληξε σε περίπου 80 λεπτομεριακά ερωτήματα τα οποία μπορούσαν να έχουν διαφορετικές ερμηνείες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η οδηγία όπως έχει διατυπωθεί θα οδηγήσει σε ασφάλεια δικαίου με τη μορφή αυτή, επομένως δεν θα φέρει κανένα πλεονέκτημα για τους πολίτες, για τις απονέμουσες αρχές ή για τις επιχείρησεις. Ωραία λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Και ας περάσουμε τώρα δεύτερο τομέα που θα μας απασχολήσει τι καθεστώς ε, θέλουμε και αν θα πρέπει αυτό να είναι ήπιο. Έχουμε άλλους τρεις ομιλητές και θα έχουν ε, όλοι από 10 λεπτά για να κάνουν τις παρουσιάσεις τους και μετά θα έχουμε ερωτήσεις από τους βουλευτές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλωσορίζω τον κύριο Μάρτιν Βέιαντ, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής για το θέμα για την υδροδότηση και τα απόβλητα, μέλος εκτελεστικού συμβουλίου, διευθυντικού συμβουλίου, του Γερμανικής Ένωσης για την ηλεκτρική ενέργεια και την διαχείριση των υδάτων. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας προοπτική για αυτή την πρόταση. 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Κατά πρώτον, κάποια επιχειρήματα νομικής φύσης. Από τη δική μου την σκοπιά, η οδηγία αυτή για τις συμβάσεις εκόρησης δεν χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα λόγω πρωτογενούς νομοθεσία και επειδή το ΔΕΚ με την ομολογία του είναι πλήρως επαρκέ ε, ως υλικό. Έπειτα, ε, οι συμβάσεις εκχώρησης δεν θα έπρεπε να εμπιπτούν στο κοινοτικό δίκαιο και δεν μπορούν να συγκριθούν με τις δημόσιε συμβάσει και του δημόσιου διαγωνισμού. Αρκούν οι κανόνε του πρωτογενού δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε τον ορισμό των όσων χρησιμοποιούνται ω τώρα, βλέπουμε ότι η σύμβαση τύπου που χρησιμοποιείται, τύπος που χρησιμοποιείται για την υδροδότηση, ουσιαστικά το σημαντικό είναι να συλλέγονται πληρωμέ για το όνομα ενό φορέα και από το λογαριασμό των χρηστών. Άρα, είναι πολύ συγκεκριμένη η κατάσταση σε σχέση με τις συμβάσεις αυτές και βεβαίως διαφέρει τελείως από τις, ε, τους δημόσιους διαγωνισμούς. Η οδηγία αυτή αναζητά ε, μια τέλεια δομή, αλλά δεν την επιτυγχάνει. Κυρίως με την ιδιωτική συμμετοχή. Στο άρθρο 15.5, αυτό που λέγεται για την ιδιωτική συμμετοχή ή την, ε, μπορεί να θεωρηθεί ως ρήτρα αποκλεισμού. Για την υδροδότηση τώρα στην ε, Γερμανία, τι μπορούμε να πούμε. Ότι είναι μια δημόσια υπηρεσία κοινοφελής. Η διαχείριση των αποβλήτων, επεξεργασία των αποβλήτων και ιδρυοδότηση εμπίπτει στη γερμανική νομοθεσία και στο δίκαιο ανταγωνισμού και είναι αρμοδιότητα των ομοσπονδιακών κατηδίων στη Γερμανία. Όπως όμως ορίζεται από την νομοθεσία ε, του άρθρου 8 του βασικού του πρωτογενούς γερμανικού δικαίου και του συντάγματο και βεβαίω και από την Ευρωπαϊκή, τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άρθρο 4. Πρέπει να διασφαλίζεται ποιότητα και αηφορία και αυτά για την υδροδότηση. Αυτό υπόκειται στη διακριτική ευχαίρεια των τοπικών αρχών να διαλέξουν την μορφή παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τώρα μια συνοπτική εικόνα των ε, διευθυντικών προποθέσεων για την υδροδότηση στη Γερμανία. Το γράφημα σας δείχνει τη μεγάλη ποικιλία του είδους επιχειρήσεων που στο επίπεδο των δημοτικών αρχών συμμετέχουν στην υδροδότηση. Διαφορετική διάρθρωση στις διαφορετικές επαρχίες της Γερμανίας. Αυτό εξηγείται επειδή υπήρξε και η πανένωση της Γερμανίας. Ε, ο βασικός στόχος ήταν η επεξεργασία του ύδατος να, εξασφαλίζει, να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα του καταναλωμένου νερού. Ε, υπήρξαν συμβάσεις που ορίζονται από την πρωτογενή νομοθεσία, οπότε οι διαρθρωτικές αλλαγές μεταξύ των κρατών μελών απαιτούν μελέτη αντικτύπου για τις διαφορετικέ συνέπειες που θα υπάρξουν. Για τη Γερμανία μπορούμε να προβλέψουμε ότι με τη συμμετοχή, τον ανταγωνισμό τέλο πάντων για την παροχή, θα μειωθούν ε, ουσιαστικά οι θετικέ συνέπειε, κάτι που είναι ο αντίθετο σκοπό από τον επιδιακόμενο τη οδηγία. Τώρα, η πρόταση για τι εκχωρήσει. Τι συνέπειε μπορεί να έχει. Η ανάθεση των συμβάσεων εκχώρηση πολλέ φορέ είναι περίπλοκη και επαχθής λόγω της προετοιμασίας της διαδικασίας διαγωνισμού που μπορεί να είναι χρονοβόρα και με περίπλοκους κανόνες και με μεγάλο κόστος επίσης, συμβουλευτικό. Η αυστηρή διαδικασία απονομής μπορεί πραγματικά να είναι υπερβολικού, υπέρμετρου άθους, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις αρχές και τους φορείς και δυσανάλογη σε σχέση με το επιδιωκόμενο εισόδημα. Αυτό στη Γερμανία με την, για την υδροδότηση είδαμε ότι υπάρχει περιφερειακή δομή και διάρθρωση σε, σε επίπεδο δημοτικών αρχών, οπότε είναι πολλές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται. Εδώ περίπου 6.000 ε, μονάδες παροχής και 8.000 για τη διαχείριση αποβλήτων συνολικά στη χώρα. Αυτά μπορεί να επηρεαστούν. Ε, το αποτέλεσμα είναι βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον ότι η πρωτογενής ε, νομοθεσία επαρκεί. Η μελέτη αντικτύπου που είδαμε ως τώρα δεν εξηγεί γιατί είναι απαραίτητη αυτή η οδηγία. Υπάρχει ανάγκη για μια νέα ε, μελέτη αντικτύπου που να μελετά την κατάσταση στα κατημέλια και τις διαφορετικές ε, συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν. Επίσης και η πρακτική κατάσταση για τι αναθέτουσε αρχέ πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώ και οι ενδεχόμενε εξελίξει στον τομέα τη υδροδότηση ιδίω. Οι κανόνε που αυτή τη στιγμή προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, αρμόζουν ούτε για την άρση τη ε, ανασφάλεια δικαίου, που, της φέληψης δικαίου που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε θα υπάρχει αυτόνομη διαδικασία λήψη αποφάσεων από τι δημοτικέ αρχέ και του φορεί τοπική αυτοδιοίκηση. Ο τομέα εντροδότηση λοιπόν ε, διζητά να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστούμε για την σαφέστατη αυτή τοποθέτηση. Θα τη συζητήσουμε ευθύ αμέσω. Επόμενο ομιλητή. Ο τομέα στον οποίο εργάζεται αναφέρθηκε προηγουμένω για λιμένες. Ο Πάτρικ Φερχόφεν είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαϊκών Λιμένων. Του δίνω λοιπόν το λόγο για 10 λεπτά. Thank you, uh, Good... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη χαρά η παρουσία μου εδώ για την παρουσίαση των απόψεων της βιομηχανίας των λιμένων και ιδιαίτερα της διαχείρισής τους. Θα ήθελα κυρίως να πω τέσσερα πράγματα. Πρώτον, να σας πω πώς χορηγούνται τα συμβόλαια μεταξύ λιμενικών αρχών και χριστών. Και έπειτα θα επισέλθω στις λεπτομέρειες των αναγκών του τομέα. Θα μιλήσω για διαφάνεια και για την απαραίτητη συνέχεια των επενδύσεων σε σύγκριση όλα αυτά σε σχέση με την πρόταση οδηγίας που έχουμε μπροστά μας. Πρώτα όμως να δούμε πώς οργανώνεται ο λιμενικός τομέας. Ιδιαίτερα τις σχέσεις μεταξύ λιμενικών αρχών που διαχειρίζονται τους λιμένες. Οι περισσότερες από αυτές είναι δημόσιες αρχές, αν και υπάρχουν και τελείως ιδιωτικές ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην υπηρετική Ευρώπη υπάρχει ένα μείγμα και δημοσίων και ιδιωτικών λιμενικών αρχών. Αυτά η οδηγία τα λέει συμβαλόμενες οντότητες, συμβαλόμενα μέρη. Με τις εταιρείες εννοείται που διαχειρίζονται το εμπόρευμα προς φορτοεκφόρτωση. Αλλά υπάρχουν και υπηρεσίες που διαχειρίζονται την κίνηση των επιβατών και επιβατριών καθώς και αποθήκευσης. Υπάρχουν και άλλων ειδών υπηρεσίες στα λιμάνια. Πολλά συμβόλαια λιμένων αφορούν και τη χρήση της γης με πολύ διαφορετικά καθεστώτα ανάλογα με τις χώρες. Σε μερικές χώρες είναι δημοσίου δικαίου, σε άλλες ιδιωτικού και στις περισσότερες μόνο ιδιωτικού δικαίου. Εκεί γίνεται μια χρήση εκτισία ανάλογα με το συμβόλαιο. Τώρα η διαφάνεια. Για μας το σημαντικό είναι να υπάρχει ευελιξία να καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής ανάλογα με την εμπορική στρατηγική μας και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο τομέας είναι πολύ δυναμικός και συμβαίνουν πολλές και ταχείες αλλαγές εκεί. Για μας λοιπόν η διαφάνεια είναι κάτι που το υποστηρίζουμε φυσικά, πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να είναι αναλογική δηλαδή. Καταρχήν να συνδέεται με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεν μιλάμε για συμβόλια που δεν όπου δεν χορηγούνται υπηρεσίες σε τρίτους, αλλάζει το πράγμα η διάρκεια του συμβολέου επίσης πρέπει να σχετίζεται το συμβόλαιο με την ε, αναμενόμενη απόδοση και υπάρχει και ο υπολογισμός του κινδύνου. Έπειτα, γενικότερα οι χωρίσεις αυτές πρέπει να θεωρούνται ως εργαλεία διακυβέρνησης, governance των λιμενικών αρχών με σύμφωνα βέβαια με τις αρχές της βιωσιμότητας, τον ανταγωνισμό και όλα αυτά. Ως προς τις διαδικασίες επιλογής εννοούμε και διαγωνισμούς και πλειονο... και γενικότερα τους κανόνες των προμηθειών. Το 28% των χωρών χρησιμοποιούν δημόσια αποκλειστικά διαδικασία, 21% μόνο εάν η γη έχει στρατηγική σημασία και 19% για άλλους λόγους και με άλλες διαδικασίες ανάλογα με τη διάρκεια του συμβολέου κτλ. Και 28% δεν χρησιμοποιούν ποτέ δημόσιες προμήθειες. Είναι κυρίως μικροί λιμένες όπου είναι χαμηλότερες οι δυνατότητες επένδυσης. Τώρα το θέμα της πρόσβασης στην αγορά και της συνέχεια των επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια ενός συμβολέου οι χρήστες του χρειάζεται να προσαρμόζονται στις αλλαγές της εσωτερικής αγοράς και εμείς ως λιμενική αρχή πρέπει να προσέχουμε να μην είναι αυτό αυτόματο δικαίωμα αλλά να δίνεται η δυνατότητα για τις εταιρείες που έχουν καλά αποτελέσματα να μπορούν να συνεχίσουν να έχουν την επιλογή να παρατείνουν το συμβόλαιό τους προτιμησιακός. Αλλιώς θα πάβουν τις επενδύσεις οι χρήστες, οι συμβολεούχοι μόλις λήξει το συμβόλαιο και έτσι θα υπάρχει χαμηλότερη αποτελεσματικότητα και λιγότερο αποτελεσματική χρήση της γης του λιμένος θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να δούμε πώς βλέπουμε το μέλλον της επένδυσης στο σε ένα υπάρχον συμβόλαιο και να δούμε αν μπορούμε να καθορίσουμε αντικειμενικές παραμέτρους ή όχι για την παράταση ενός συμβολέου. Τέλος, ορισμένα σε πιο συγκεκριμένα θέματα της οδηγίας, κάναμε πολλές συζητήσεις με την Κομισιόν γιατί στη Γενική Διεύθυνση Αγορών και ευχαριστώ την Γενική Διευθύντρια για τις συζητήσεις αυτές. Για μας η αξία της οδηγίας αυτής ακόμη συζητιέται. Είναι συζητήσιμη. Υπάρχει βέβαια το θετικό στοιχείο να υπάρξει ένα γενικό κοινό πλαίσιο για τη διαχείριση των λιμένων για να υπάρχει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα, αλλά ένα από τα κυριότερα θέματα που συζητάμε είναι το εύρος της, γιατί η χορήγηση εκχωρήσεων συμβολέων για λιμένες δεν μπορεί να γίνεται αυτόματα, δεν είναι όλες οι προσφορές κατάλληλες. Είναι φανερό ότι συμβόλαια που προβλέπουν και υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος όπως την εκπαίδευση πιλότων κλπ. Για μας είναι πιο ενδιαφέρον τα συμβόλαια αυτά από τα υπόλοιπα που δεν περιέχουν τέτοιες ρήτρε. Προς στιγμή λοιπόν προβλέπουμε την πρόταση να προτείνουμε και συμπληρωματικό εργαλείο τρία θέματα κυρίως μας ενδιαφέρουν Δηλαδή το όριο, τα 5 εκατομμύρια που για μας είναι πολύ χαμηλό, γιατί συμπεριλαμβάνει σχεδόν όλα τα συμβόλαια, άρα για μας χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι δύσκολο να οριστεί το όριο σε μια οριζόντια οδηγία, ίσως το κριτήριο να είναι η επιφάνεια του λιμανιού ή άλλο κριτήριο. Επίσης τα διαδικαστικά που χρειάζονται εδώ που προβλέπει η οδηγία για μας είναι υπερβολικά αυστηρά και καταστρέφουν τη δυναμικότητα του τομέα. Ιδίως όταν μιλάμε για πιθανές τροποποιήσεις και παρατάσεις των συμβολέων που για μας είναι ουσιαστικό θέμα και δεν το αναφέρει ρητά η οδηγία. Τα περισσότερα από αυτά με χαρά διαπίστωσα ότι στην πρώτη χρωμοδότηση του εισηγητή ελήφθησαν υπόψη. και η τελική μας αξιολόγηση της οδηγίας θα εξαρτηθεί από τις τροπολογίες που θα κατατεθούν στο Κοινοβούλιο και το Συνεβούλιο. Σας κατευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη σαφήνεια των απόψεών σας και των θέσεών σας. Ο τελευταίος και λουκούμιος ομιλητής μας είναι ο Στεφάν Σεσχέ, ο οποίος είναι καθηγητής στην επιχειρηματική σχολή της ε, Σορβόνης όπου κάνει ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τις εταιρικέ σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Για 10 λεπτά λοιπόν έχετε το λόγο σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Ως τελευταίος ομιλητής θα ήθελα να αναφέρω ορισμένες σκέψεις ως πανεπιστημιακός. Δεν είμαι εδώ για να υποστηρίξω ένα βιομηχανικό κλάδο ή μια, κάποια επιχειρηματικά συμβόλαια και θέσεις, αλλά να αντιμετωπίσω από επιστημονική και ερευνητική άποψη τα θέματα αυτά των δημοσίων συμβάσεων και γι' αυτό θέλω να δώσω τις απόψεις μου για τα στοιχεία αυτής της οδηγίας που φαίνεται ότι είναι λογικά και αυτά τα οποία είναι βελτιώσιμα από την άλλη πλευρά. Πρώτα απ' όλα, γιατί χρειάζεται να υπάρξει ένα νέο καθεστώς το οποίο να διέπει τις συμβάσεις εκχωρήσεων, ιδίως εκχωρήσεων υπηρεσιών. Η οδηγία που συζητείται σήμερα μου φαίνεται ένας καλός τρόπος να επιτευχθεί ο στόχος της μεγαλύτερης διαφάνειας και της σαφήνεια σε σχέση με τους δημόσιους διαγωνισμούς εκχωρήσεων, ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ασάφεια και να μην υπάρχει τόσο μεγάλο περιθώριο επιλογής για τις αρχές απονομής, να υπάρχουν σαφείς κανόνες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πιο εύκολα οι φορεί τους διαγωνισμούς. Από την άποψη αυτή, αυτή η προσπάθεια που γίνεται με την οδηγία αυτή να γίνουν πιο διάφανε οι συνθήκες, δυνητικά θα βοηθούσε τον ανταγωνισμό. Και συμφωνώ με τον Μάικλ Μπρουνέτ για το θέμα αυτό. <clears throat> το πραγματικό ερώτημα όμως, το οποίο προκύπτει και από τις ε, παρεμβάσεις και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα, είναι γιατί χρειαζόμαστε ένα ελαφρό καθεστώς ή θα ήταν καλύτερο να έχουμε ένα πιο ε, συγκροτημένο πλαίσιο. Υπάρχει εδώ μια διαφορά μεταξύ αυτών που θέλουν μια εκτατική μορφή διαπραγματεύσεων για τις συνθήκες εκχωρήσεων και αυτών που θέλουν να υπάρξει μια ενιαία οδηγία μεταξύ των δημοσίων συμβάσεων και των εκχωρήσεων, οπότε να περιοριστεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης στην επιλογή του αναδόχου. Υπάρχουν διαφορετικές ε, απόψεις σε σχέση με την ε, ε, οικονομική βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά. Η θεωρία των ατελών συμβάσεων αντιμετωπίζει το θέμα αυτό και τονίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των συμβάσεων εκχωρήσεως. Γιατί εκεί πρόκειται <clears throat> για συμβάσεις όπου πολύ συχνά υπάρχουν επεμβάσεις, ε, επενδύσει, συγγνώμη, υπάρχει μεταφορά κινδύνου, είναι μακροχρόνιες συμβάσεις και είναι πολύπλοκες ε, συμβάσεις που αφορούν πολύπλοκες δημόσιες υπηρεσίες που είναι πολύ δύσκολο για την απονέμουσα αρχή να καθορίσει ακριβώς τι περιμένει από τον ανάδοχο και είναι πολύ δύσκολο να προκαταλάβει και τις εξελίξεις μελλοντικέ στην αλλαγή των ε, αναγκών και του γούστου του καταναλωτή. Βρισκόμαστε λοιπόν σε συμβόλαια σε συμβάσεις που είναι πιο πολύπλοκα από αυτά των δημοσίων ε, συμβάσεων και επομένως υπησέρχονται στην θεωρία των ατελών συμβάσεων, των συμβάσεων που θα πρέπει να τύχουν επαναδιαπραγμάτευσης γιατί δεν μπορούν να προβλεφθούν όλα τα στοιχεία εκεί. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ακαδημαϊκή ε, βιβλιογραφία, αν θέλετε, για τα άμεσα, για τα ατελή συμβόλαια που δείχνει ότι από τη στιγμή που ξέρουμε ότι είναι πολύπλοκα αυτά τα συμβόλαια, ότι πρέπει να τύχουν αναδιαπραγμάτευσης, δεν είναι πάντα πολύ αποτελεσματικό και, πιο, και πολύ λογικό να έχουμε άκαμπτες και συγκεκριμένες ε, διαδικασίες ε, απονομής. Αντίθετα, θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη στάθμιση των κριτηρίων. Οι ερευνητικές λοιπόν Μελέτε. λένε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μα πράγματα που δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στη μελέτη, όπω είναι στην πρόταση τη Κομισιόν, όπως χάρη η εμπειρία και η εμπειρογνωμοσύνη του αναδόχου, ιδίω όταν πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αναδιαπραγμάτευση των ε, συμβολέων. Από την άποψη αυτή υπάρχουν ορισμένα στοιχεία θεωρητικά που δείχνουν ότι θα είναι καλό να αφήσουμε ανοιχτή τη δυνατότητα αναδιαπραγμάτευσης μέχρι ενός σημείου των ε, ε, συμβάσεων εκχωρήσεω, ιδίω για αυτέ οι οποίε έχουν μεγάλη πολυπλοκότητα τις συμβάσεις. Και ότι δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε πάντα κριτήρια τα οποία είναι αυστηρά και να τα σταθμίσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το δεύτερο πράγμα το οποίο γνωρίζουμε από θεωρητική άποψη και υπήρξαν πολλές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα αυτό είναι ότι στις συμβάσεις εκχωρήσεων η επαναδιαπραγμάτευση είναι ο κανόνα και όχι η εξαίρεση στις περισσότερες αυτές τις μακροχρόνιες συμβάσεις υπήρξε μια αναδιαπραγμάτευση για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές συνθήκων. Κάποιες μελέτες εδώ βλέπετε που έγιναν σε εκχωρήσεις στη Λατινική Αμερική μεταξύ του 1980 και του 2000 από την Παγκόσμια Τράπεζα που λέει ότι πάνω από 40% από αυτά τα συμβόλαια έχουν τύχει αναδιαπραγμάτευση μετά από λιγότερο από δύο χρόνια για λόγους οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι αρνητικοί λόγοι. Έχετε επίση τι εμπειρίε του Μεγάλη Βρετανία που δείχνει ότι έχει υπάρξει ένα μεγάλο αριθμό αναδιαπραγμάτευσης και αυτό γιατί έχουν ιδιαίτερα άκαμπτο χαρακτήρα. Αυτά δείχνει η έκθεση τη Βουλής των Κοινοτήτων το 2011. Έχετε τι εκχωρήσει για τα πάρκινγκ στη Γαλλία που λέει ότι κατά μέσον όρο μια, ιδιο... Κάθε δύο χρόνια περίπου γίνεται μια αναδιαπραγμάτευση και αυτό φαίνεται ότι είναι προ όφελο των καταναλωτών. Επίση, έχετε εμπειρίε στι ΗΠΑ που δείχνουν ότι γενικά ο κανόνα είναι αναδιαπραγμάτευση. Μπορεί κανεί να προχωρήσει σε αναδιαπραγμάτευση γιατί ο ανάδοχος πολλές φορές μπορεί να εξασφαλίζει τμήμα της πίτας Πολλέ φορέ γίνεται διαπραγμάτευση για λόγου διαφθορά. πολλέ φορέ όμω γίνεται διαπραγμάτευση για πραγματικού λόγου γιατί πραγματικά χρειάζεται να υπάρξει μια αναδιαπραγμάτευση και μια προσαρμογή στι νέε συνθήκε. Για αυτά θέλω να τονίσω από τι οικονομικέ αυτέ μελέτε προκύπτει η έννοια ότι τα συμβόλαια αυτά έχουν ένα ειδικό χαρακτήρα και πρέπει να παραμείνει και κάποιο περιθώριο για τις απονέμουσες αρχές σε ό,τι αφορά την επιλογή των εταίρων και σε ό,τι αφορά τις δυνατότητε αναδιαπραγμάτευσης. Σίγουρα όμως χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια για να αποφύγουμε τις καταχρήσεις στον τομέα αυτό. Να εξασφαλίσουμε ότι έχει αιτιολογηθεί πλήρως η επιλογή της δημόσιας αρχές σε σχέση με τον ανάδοχο και την αναδιαπραγμάτευση ότι να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι θετικού αθρίσματος, ότι κερδίζει και ο ανάδοχος και η, η τοπική κοινότητα και οι δημόσιες αρχές. Και όλα αυτά με οδηγούν σε ορισμένα συμπεράσματα ότι το να έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό στις συμβάσεις εκχωρήσεων δεν είναι δωρεάν γεύμα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις. Θα μπορούσε να γίνεται μονάχα αν υπάρχει μια αρχή η οποία είναι σε θέση να κάνει ένα τέλειο έλεγχο όλων αυτών των στοιχείων που προανέφερα και αυτό από ό,τι γνωρίζω δεν προβλέπεται από την οδηγία. Έχω μόνο δύο λεπτά, θα πάω πολύ γρήγορα, θέλω να τονίσω ότι η οδηγία αυτή πλησιάζει τον ε, νόμο Σαπτά, ο οποίος ισχύει στη Γαλλία από το 1993. Ο νόμος αυτός, για να σας τον παρουσιάσω με απλό τρόπο, είναι σαν τη σημερινή οδηγία, πιο απλός, λιγότερο δεσμευτικός. Η εμπειρία μας είναι ανάμεικτη προστοθετική από την άποψη ότι έχει μειωθεί κατά 8% για τον καταναλωτή η, το τίμημα των συμβάσεων. Στις μεγάλες πόλεις έχει φτάσει και στο 15%. Αυτό δείχνει ότι έχουν μεγαλύτερη διαπραγματική ικανότητα στις μεγάλες πόλεις. Αλλά από την άλλη μεριά ο αριθμός των προσφορών είναι ε, σχετικά μικρός. Και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον για την οδηγία είναι ότι αυτό το οποίο επιζητεί είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ε, δυνητικών προσφορών και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Κλείνω λοιπόν τονίζοντας ότι κατά την άποψή μου είναι απαραίτητο η οδηγία αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή διότι ο διάβολος διαμένει μεταξύ των λεπτομεριών όπως γνωρίζουμε και παραδείγματος χάρη θα πρέπει η διάρκεια <clears throat> μιας ε, σύμβασης να μην βασίζεται μονάχα στις ε, επενδύσεις αλλά και στους επιδιωκόμενους στόχους, στην μεταφορά κινδύνου κτλ. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για τον ορισμό των συμβάσεων εκχωρήσεως και τη μεταφορά του κινδύνου και αναρωτιέμαι μήπως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις καινοτομίε στο συμβατικό δίκαιο που βλέπουμε στις συμβάσεις εκχωρήσεως, δηλαδή συμβάσεις που έχουν μακρόχρονικό διάστημα, αλλά που πράγματι διακόπτονται τα σε ένα ορισμένο επίπεδο ο τζίρος του αναδόχου, επομένως θεωρείται ότι ο κίνδυνος έχει καλυφθεί. Επίσης, το θέμα του, της εξαιρέσεως ορισμένων προσφορών που θεωρούνται πολύ χαμηλές και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αποκλείσουμε ε, υποψηφιότητες που έχουν δείξει στο παρελθόν μια στάση διαφθοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, αναπληρωτά καθηγητή. για την παρουσίασή σας και που συμπεριλάβετε τόσα πολλά στοιχεία. Ήταν πολύ πλούσια. Αρχίζει τώρα η συζήτηση με τον εισηγητή και τους κοιόδους εισηγητές. Θα καλέσω πάλι πρώτα τον κύριο Ζήβα να κάνει τα σχόλιά του και μετά τους συναδέλφους. Αλλά θα τους παρακαλέσω να παραμείνουν στο δίλεπτο. Θέλουμε να έχουμε λίγο χρόνο και για την κυρία Σικόφσκα. Κυρία Ζουβά. Η κυρία Βερνιό, η κυρία Ρούλε, ο κύριος Μπερνόε. ο κύριος Παντζέρη, η κυρία Κέπχαρτ, κυρία Βάιλερ, κυρία Φανχέρεν. Oh. Uh, so Άλλος κανείς Δύο λεπτά ο καθένα περίπου, παρακαλώ, ώστε να προλάβουμε να ακούσουμε και τι απαντήσει. Εάν μείνετε και σε λιγότερο από δύο λεπτά, τόσο το καλύτερο. Κύριε Ζουβά. Mr. Mr. Panzeri, Mr. Mrs. Uh, uh, then others. Uh, και λυπή. Κύριε Ζουβά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα πρώτο ερώτημα για το μη πλήρες συμβόλαιο μιλήσατε. Μπορείτε να μας σχολιάσετε ποια ακριβώς αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαφάνεια γιατί δεν ήταν διαφανές αυτό που είπατε. Δεύτερη παρατήρηση προς τον κύριο Βεγιάντα. Βρίσκω ειλικρινά ότι το να λέτε και να γράφετε ότι λόγω του πρότασης αυτής δεν υπάρχει πια αυτονομία στη λήψη αποφάσεων από τις τοπικές αρχές είναι απλώς ανακριβές. Μπορείτε να πει, μιλήστε υπέρ, κατά, αποχές, αλλά δεν μπορείτε να το πείτε αυτό. Σε κανένα σημείο του κειμένου δεν γράφει ότι οι τοπικές αρχές χάνουν την αυτονομία της λήψης αποφάσεών τους, αφού αυτές μπορούν να αποφασίσουν τελείως ελεύθερα να δεχτούν ή όχι μία εκχώρηση. Δεν βλέπω λοιπόν πού, σε ποιο σημείο, σε ποιο άρθρο μειώνεται η αυτονομία της λήψης αποφάσεων των τοπικών αρχών. Σας τα λέω με εκνευρισμό διότι τέτοιου είδους κείμενα διατρέχουν τον κίνδυνο να επικριθούν ε, αδίκως για πράγματα που δεν τα γράφει μέσα. Ερωτώ λοιπόν, πού το λέει. Δεύτερον, όταν λέτε ότι δεν χρειάζεται νομοθεσία διότι υπάρχει η νομολογία, εμείς είμαστε βουλευτές και σε δημοκρατία δεν κρίνει ο δικαστής. κάτι που βγαίνει από την ομολογία δεν μας ικανοποιεί. Κάθε δύο χρόνια περίπου βγαίνει μια δικαστική απόφαση για μια συγκεκριμένη εκχώρηση, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί βάση για λήψη αποφάσεων. Εγώ προτιμώ κανόνες που να τους ορίζει δημοκρατικά το κοινοβούλιο. Όχι κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια να αλλάζει ανάλογα με τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ορίστε, αυτά. Ευχαριστούμε ο κύριος Παντζάλη. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τον Τζουβέν με αυτά που είπε. Όντως, εδώ ακούμε πυρογνώμονες, τεχνικούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να αποφασίσουμε από πολιτικής άποψης και ως νομοθέτες. Όμως, Νομίζω η νομοθετική επιλογή είναι σκόπιμη. Σκοπό έχει να προωθήσει και τις εκχωρήσεις και να υπάρχει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των συμβάσεων. Εδώ λοιπόν, ακούγοντας τους προσκεκλημένους μας, καταλαβαίνω ότι είναι σαφές. Χρειαζόμαστε έναν ορισμό πιο σαφή για τις εκχωρήσεις. Κάτι ανάλογο με τις διατάξεις για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Υπάρχουν βεβαίως έννοιες που είναι πολύ ε, συγκεκριμένες και τις οποίες θα πρέπει να δούμε με ευελιξία γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ δημοσίων συμβάσεων και εκχωρήσεων. Για τη διαδικασία των διαγωνισμών πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο διαλλακτικό, ευέλικτο, που να μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό. Νομίζω λοιπόν σκόπιμο είναι να είναι διαφανέστερο αυτό το πλαίσιο της ουσίας να μην επιτρέπει διακριτική μεταχείριση ούτε την παράβαση των δικαιωμάτων των δημοσίων αρχών. Να έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται με βάση τη διακριτική τους ευχέρεια και να ανοίγουν στην ανταγωνιστικότητα και στον ανταγωνισμό την παροχή κάποιων υπηρεσιών. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει αναγνώριση της δυνατότητας αυτοοργάνωσης και αυτοδιοργάνωσης των δημοσίων αρχών σε σχέση με τις εκχωρήσεις. Τώρα ερωτήσεις. Είναι απαραίτητο και αυτή την παρατήρηση θέλω να την κάνω τόσο ή άλλως για να ακούσω και τα σχόλιά σας. Είναι απαραίτητο να ορίσουμε καλύτερα τα κριτήρια των εκχωρήσεων λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο ένα θέμα που επανελειμμένως αναφέρθηκε, την διάρκεια των επενδύσεων, αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να δούμε εντό εισαγωγικών τις παραδόσεις που ισχύουν στα διάφορα κατημέλη. ώστε να ξέρουμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη και σε αυτόν που ανέλαβε το έργο. Και έπειτα τελευταία παρατήρηση για τις in-house υπηρεσίες. Εδώ υπάρχει μια ενιαία αγορά και είναι σαφές ότι ο δημόσιος φορέας θα πρέπει να κάνει κάποια επιλογή. Αλλά μπορεί να μην υπάρχει ανάλογη αγορά υπηρεσιών. Εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα ερώτημα. Τι πρέπει να γίνει μπορούμε να αφήσουμε τον χώρο να καλυφθεί από το δημόσιο τομέα ή να υπάρξει ένα καθεστώς ανταγωνιστικό, δηλαδή άνοιγμα της αγοράς. Οι επιλογές αυτές θα πρέπει να γίνουν και μάλιστα συγκεκριμένα. Ακριβώς γιατί υπάρχει απέτηση να υπάρχει ένα διαφανές και σαφές νομοθετικό πλαίσιο. Ε, Ευχαριστούμε, συνάδελφοι. Παρακαλώ να επικεντρώνεστε σε ερωτήσεις, εφόσον έχουμε εδώ και τους και Κύριε Μπουζόη. Ευχαριστώ. Δεν θα ξεπεράσω τα δύο λεπτά. Είναι σαφέ αφού άκουσα αυτές τις εξαιρετικέ παρουσιάσεις, ότι θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά. Όχι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε σωστά τη δουλειά της, εξαιρετικά την έκανε, αλλά έχουμε εδώ ένα θέμα περίπλοκο να αντιμετωπίσουμε με πολλές λεπτομέρειες και πολλέ ε, ιδιαίτερες περιπτώσεις ανάλογα με τον τομέα. Βλέπουμε άλλες ανάγκες να αναφέρονται από την Ένωση Βιομηχάνων ή από την ε, Ένωση Λιμένων. Πρέπει λοιπόν προφανώ να βρούμε και τις ανάλογες λύσεις. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε κατά πρώτον τον ορισμό των εκχωρήσεων. Είναι καθοριστική σημασία προκειμένου να διευκολύνουμε την διάκριση, μεταξύ δημοσίων συμβάσεων, εκχωρήσεων, εκχωρήσεων έργων και εκχωρήσεων υπηρεσιών. Δεν συμφωνώ με τη δήλωση ότι δεν χρειαζόμαστε την οδηγία, διότι έχουμε πλέον κατακαιρματισμό, ε, έλλειψη διαφάνεια και έλλειψη ικανοποίηση των ε, ενδιαφερομένων. Η κατάσταση που ισχύει λοιπόν σήμερα δεν είναι σε καμία περίπτωση ιδανική. Πρέπει να συμφωνήσω με όσους επέκριναν την μελέτη αντικτύπου ήταν ε, ελλειπής. Δεν κάλυψε όλα τα ζητήματα ή όλες τις περιπτώσεις που μας απασχολούν. Αυτό κάνει τη δουλειά μας λίγο πιο δύσκολη. Έχω μια ερώτηση για τη διάρκεια. Είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ διάρκειας, που ε, έχει να κάνει βεβαίως και με την ε, απόσβεση των επενδύσεων, και με τον οικονομικό κίνδυνο που είναι ε, ένα στοιχείο γενέ των εκχωρήσεων. Πώ μπορεί αυτό να καθορίσει τα χαρακτηριστικά των εκχωρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που παραμείνετε μέσα στα δύο λεπτά σα, κυρία Ρούλα, για δύο λεπτά. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στον κύριο Ζουβέν. Λέτε ότι πολλέ διαδικασίε έχουμε στον τομέα αυτό. Πρέπει να σκεφτείτε ότι έχουμε πολύ περισσότερες υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις και αυτό δεν έχει οδηγήσει, τα 40 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν οδηγήσει στο να μειωθούν αυτές οι διαδικασίες. Είναι αμφισβητήσιμο λοιπόν ότι ξέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιο τρόπο που θα μειώσει τις προσφυγές. Θα ήθελα σταθώ στην τελευταία παρουσίαση γιατί είπατε αν κατάλαβα καλά είναι διαφορετικό το είδος των συμβάσεων εδώ από ότι στις ε, δημόσιες συμβάσεις. Είναι διαφορετικές, είναι ατελείς λοιπόν συμβάσεις οι οποίες απαιτούν μια μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Και τότε θέλω να θέσω ένα ερώτημα, εάν ισχύει αυτό που είπατε. Ο πρώτος ομιλητής είπε ότι θα μπορούσαν οι συμβάσεις εκχωρήσεων για υπηρεσίε να συμπεριληφθούν στις δημόσιες συμβάσεις. Εσείς είπατε όχι, ότι είναι τελείω διαφορετικό. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε αν πιστεύετε πράγματι ότι μπορούν να συμπεριληφθούν στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις εκχωρήσεων. Εγώ πιστεύω και εγώ ότι είναι διαφορετικού χαρακτήρα. Ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν κατάλαβα καλά, συμφωνείτε όλοι ότι η πρόταση Κομισιόν είναι ιδιαίτερα πεπλεγμένη και δεν είναι στο ύψος των αναγκών. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αναδιαμορφώσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σας για το θέμα αυτό, γιατί αυτό τότε δεν, η πρόταση Κομισιόν δεν ανταποκρίνεται στην έκθεση επιπτώσεων που αναφέρθηκε και θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος ε, Ζουβέρ για το θέμα της διαφάνειας που είναι κεφαλαίωδης για τις συμβάσεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα σε εταιρικό επίπεδο. Και ίσως και η, η αναθεώρηση των συμβάσεων αυτών θα πρέπει να καλύπτεται από περισσότερη διαφάνεια και όχι μονάχα η αρχική σύμβαση. Νομίζω ότι η κύρια επίκριση η οποία ε, ισχύει για τις συμβάσεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία και ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά εξάλλου είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια. Ωραία, λέει ο κύριος Χάμπορ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε να ψηφίσουμε στις 11 και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη της Κομισιόν και να απαντήσουν και οι εμπείρο Η κυρία Βανιού Μπερναδέτη. Βεβαίω θα είμαι πάρα πολύ σύντομη κύριε Πρόεδρε, διότι το θέμα αυτό το οποίο ήθελα να δείξω είχε καλυφθεί και από τον εισηγητή. Αναφέρομαι στον κύριο Σουσί, μιλήσατε για win-win-win, για θετικό άθροισμα και περιπλέον. Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει τώρα με, την, ε, με τις δημόσιες ιδιωτικές εταιρικές σχέσεις και δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τον καταναλωτή. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα πρόσθετο φορέα. Αυτό μου φαίνεται ενδιαφέρον. Τι πιστεύετε όμως για την δομή αυτού του πρόσθετου φορέα, ποιες θα είναι οι αποστολές που θα πρέπει να φέρει σε πέρας και θέλω, είμαι πάρα πολύ σύντομη όπως βλέπετε, να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και η ακρόαση, ακόμα και αν έχω μείνει με περισσότερα ερωτήματα από απαντήσεις στο τέλος της συζήτησης. Και εγώ σύμφωνα μαζί σας. Αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ καλή ακρόαση. Λοιπόν, να σας πω ποιος ακόμα είναι στον κατάλογο. Βάιλε, Μαχέβα και Γκέπχαρτ. Άλλος. Α, και ο κύριος ε, Σουάμπ, βεβαίως. Γεια. Παρακαλώ, αν μπορείτε να παραμείνετε σε επίπεδο συντομία, πρώτη η κυρία Βάιλα. Γεια, ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση για το θέμα που έθεξε ο κύριος ε, Ζουβέν και η κυρία Ρούλα. Είναι το θέμα της ασφάλειας δικαίου και οι πολλαπλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα θέματα αυτά. Εγώ θα χαιρόμουν αγαπητοί συνάδελφοι αν έφτανε το πρωτογενές δίκαιο στον τομέα αυτό. Δεν είναι η εντύπωσή μου όμως ότι επαρκεί. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Πολλές φορές το δίκαιο των συμβάσεων δεν λαμβάνεται υπόψη επαρκώς το δικαίωμα του ανταγωνισμού. Αλλά για τις ε, Συμβάσει εκχωρήσεω είναι διαφορετικές οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι σημαντικές και είναι διαφορετικές. Ακριβώς γι' αυτό χρειαζόμαστε μια χωριστή οδηγία γιατί δεν επαρκεί το πρωτογενέ δίκαιο. Βλέπουμε ότι δεν συμφωνούν και αντιφάσκουν μεταξύ τους οι ομιλητές και αυτό δεν με πείθει ότι έχουμε ασφάλεια δικαίου, αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει να μην υπάρξουν μειώσεις ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών και να μην υπάρξουν ε, άσκοπες ιδιωτικοποίησεις. Στο άρθρο 15 υπάρχει μια ρήτρα ε, πρόληψης έναντι της ιδιωτικής ε, συμμετοχής σε τέτοιες διαδικασίες. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό και έρχομαι πάλι στο θέμα της ειδοδότησης. Δεν είναι ότι είναι παράδεισος για την υδροδότηση η Γερμανία πάντα έχω προβλήματα γιατί λέει η κυβέρνηση του κρατηδίου μου ότι είναι πάρα πολύ ψηλέ οι τιμές και θα πρέπει να υπάρξει ανταγωνισμός. Υπάρχουν συνέχεια καυγάδες <clears throat> και διαμάχες για τα θέματα της υδροδότησης μεταξύ δήμων και άλλων ε, αρχών. Εγώ δεν εκπροσωπώ βέβαια το κρατήριο της χέσης, αλλά με ενδιαφέρει να λειτουργούν καλά αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό εγώ δεν υποστηρίζω την αντιμετώπιση αυτή ε, να υπάρξει μια τέτοια μορφή ιδιωτικοποίησης που στο κρατήδιό μου στην ΕΣΥ εγώ δεν είδα να λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα λοιπόν να μου εξηγήσετε λίγο περισσότερο για το θέμα αυτό, γιατί και στη Γερμανία τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από ό,τι μπορεί να φαίνονται επιφανειακά. Ευχαριστώ. Κύριε Βάιντα. Η κυρία Φερχάιεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ δύο ερωτήματα. Είναι σαφές. Είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες για όλους τους φορείς που καλύπτονται από, τις διαφορε... την οδηγία αυτή και μπορεί να υπάρχουν διάφοροι κανόνες από ότι βρίσκονται απλώς στις οριζόντιες οδηγίες και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει απαραίτητη ευκαλυψία Επομένως, είναι απαραίτητο η οδηγία να λάβει υπόψη την πολυπλοκότητα στην πραγματικότητα που έχουν οι διάφορες μορφές συμβάσεων εκχώρησης, όπως ζητείται και από, τους, από τις αρμόδιες αρχές. Υπάρχουν βασικά θέματα όπως η διαφάνεια, η μη διάκριση κτλ. Αλλά πρέπει να διατηρηθεί και η ευκαμψία. Ένα ερώτημα στον κύριο Σουσιέ. Λέτε ότι η οδηγία αυτή είναι προσαρμοσμένη στο νόμο ΣΑΠΑ, το γαλλικό. Εγώ βλέπω ότι είναι πολύ πιο πολύπλοκη από αυτά που λέει ο νόμος ΣΑΠΕΝ. Είναι πιο ασφα, είναι πιο αυστηρή αυτή, η πιο αυστηρή αυτή η αντιμετώπιση είναι απαραίτητη και είναι ε, για να αντιμετωπιστούν τα θέματα των συμβάσεων που καλύπτουν διάφορες τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η κουλτούρα, το νερό, οι λιμένες, Όλα αυτά λοιπόν που έχουν να κάνουν με εκχωρήσεις, εκχωρήσεις αδειών, υπάρχουν πάρα πολλές λοιπόν ε, ε παραλλαγέ στα θέματα, παραγωγικά για ένα ιδιωτικό σχολείο, οι συμβάσει για την εκμετάλλευση κάποιου ακινήτου. Είναι τόσο πολλέ αυτέ οι μορφέ συμβάσεων, ώστε πρέπει να παραμείνει η ανάγκη τη ευκαμψία για του Δήμου και να λάβουμε υπόψη μα πάντα ότι μια άκαμπτη μορφή ρύθμισης όπως είναι παραδείγματος χάρη η πλήρης μεταφορά κινδύνου δεν είναι πραγματικά επιτεύξιμη παντού. Πώς λοιπόν βλέπετε αυτή την ε, πρόταση οδηγία συνεπαρκής. Και οι τελευταίοι ομιλητές, κύριε Γκέπχαρ και ο κύριος Σουάπ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι ένα πράγμα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφές. Ότι θα πρέπει να ε, πράξουμε ορισμένα σε αυτή την οδηγία. Ακόμα και όταν, κύριε Ζουβέν, βλέπετε ότι δεν προβλέπετε μια διαδικασία ε, ιδιωτικοποίησης, να το κάνουμε σαφές ότι δεν είναι αυτό ο στόχος αυτής της οδηγίας. Θα πρέπει να είναι σαφές τι καλύπτει αυτή η οδηγία και τι δεν καλύπτει. Ένα δεύτερο θέμα όπου πρέπει να είμαστε σαφείς είναι ο ορισμός των συμβάσεων εκχωρήσεων. Και γι' αυτό Εμεί αποφασίσαμε ω συντονιστέ τι προτάσει σα ότι θα πρέπει να ερευνήσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το θέμα, ώστε να υπάρχει σαφήνεια στις, ε, στον ορισμό των εκχωρήσεων περί τίνος πρόκειται και ποιε είναι οι περιπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται. Να μην υπάρχουν διαφορετικοί επίσης ορισμοί στην οδηγία από ό,τι στα κράτη-μέλη, γιατί αυτό δεν θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Κύριε Σωσιέ, είχα να θέσω ένα ερώτημα σε εσά ή μάλλον δύο ερωτήματα. Όταν μιλήσατε για τον νόμο Σαπέν ότι πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση με την οδηγία όπως είπε και η κυρία Φερχάιαν προηγουμένως, εσείς <clears throat> βλέπετε, είπατε ότι είναι πιο ευέλικτος ο νόμος Σαπέν από αυτά τα οποία περιλαμβάνει πρόταση της Κομισιόν, θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε αυτό καλύτερα, να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα. Και επίσης είπατε ότι τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Λόμου Σαπέμ φάνηκαν στις μεγάλες πόλεις. Μήπως μπορεί κανείς να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι αυτός ο νόμος ευνοεί τα πράγματα στην περίπτωση των μεγάλων πόλεων, των μεγάλων συμβάσεων. Μήπως αυτό λοιπόν έχει κάποια επίπτωση στα κατόφλια τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρώτη Κομισιόν. Ένα τρίτο σημείο πάρα πολύ σύντομα, στα, για να παραμείνω μέσα στα δύο λεπτά. Είπατε ότι ένα πιο ελαφρό και απλό σύστημα είναι απαραίτητο, ότι πέραν της ε, διαφάνειας θα πρέπει όλα αυτά τα άλλα στοιχεία να μην βρίσκονται στην οδηγία. Συμφωνείτε με αυτό ή όχι. Ευχαριστώ και τέλος ο κύριος Σουάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε καθηγητά Μπερνέτ, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Είμαι από τους πρώτους οι οποίοι υποστήριξαν αυτή την πρόταση και τόνισα ότι πρέπει η, η οδηγία για τις εκχωρήσεις να συμπεριληφθεί πλήρως στην οδηγία στη λογική των δημόσιων συμβάσεων. Εσείς υποστηρίξατε και εσείς αυτή τη θέση. Το ερώτημά μου είναι σε σχέση με την έκθεση επιπτώσεων. Υπάρχει ένα ερώτημα, υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν απαντηθήκαν μεταξύ των οποίων και οι ορισμοί. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Θα οδηγήσει αυτή η πρόταση στο να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατότητα χρήση του μοντέλου ιδιωτικών δημοσίων εταιρικών σχέσεων σε επίπεδο Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίση θα βοηθήσει σε τομείς όπως ε, είναι παραγωγικά, χάρη υδροδότηση και άλλοι, να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις. Δηλαδή υπάρχουν οικονομικά ωφέλη τα οποία θα προκύψουν από αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλατε ο κύριος Μπερνέτ να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Εντάξει, θα του δώσω το λόγο στο τέλος. για να μην νιώθουν ε, ότι αποκλείονται οι άλλοι εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει όλοι να έχουν ένα σύντομο διάστημα για να απαντήσουν αν θέλουν. Δεν κάνω διακρίσει λοιπόν και αυτό είναι ένα από τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Αν έχω και εγώ λίγα δευτερόλεπτα. Είχαμε πολλές συζητήσεις για την ασφάλεια δικαίου. Ο κύριος Σούση στην παρουσίασή του τόνισε ιδιαίτερα το θέμα της ε, των εκχωρήσεων, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις καθορίσει κανείς με ένα ορισμό γιατί είναι τόσο πολύμορφες. Και ανέφερε ο κ. Σούση ότι λόγω της πολυπλ... πολυπλοκότητας τους η αναδιαπραγμάτευση είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Τούτου λεχθέντος. Ναι. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά στη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Αλλά το θέμα της απονομής και αυτό που λέει ο κ. Μπερνέτ, τα κριτήρια απονομής και ανάγκη διαφάνειας και ανοιχτού ανταγωνισμού. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι κοινό σε όλο το φάσμα των δημοσίων προμηθειών και αγορών. Και αυτή είναι ίσως η ισορροπία που θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο σε όλους τους ομιλητές στη δεύτερη ε, γύρα. Θα δώσω τον κύριο Σωσία, τον κύριο Φερχέν και στον ε, άλλο ομιλητή το χρόνο για να απαντήσουν και δεν ξέρω αν και οι άλλοι τρεις ομιλητές θέλουν να απαντήσουν. Όχι σίγουρα ο κ. πρέπει να απαντήσει το ερώτημα του κ. Σουάπ. Καθηγητές Σοσιέ. Ε, Πραγματικά είναι challenge να απαντήσω σε δύο λεπτά. Σε οκτώ ή εννέα ερωτήσει που σημείωσα. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικό. Σε ό,τι αφορά την αρχή που θα μπορούσε να εξασφαλίζει περισσότερη διαφάνεια ναι, θα ήταν μια κατάσταση win-win-win εάν συνέβαινε. Έχουμε αριθμούς και στατιστικά στοιχεία που δείχνει ότι οι επαναπληρωματεύσει οδηγούν σε διαφορετικέ ερμηνείε. Τελικά διαπραγματευόμαστε για του σωστού ή του λάθο λόγου. Και δεν πρέπει να υπάρχουν αρχέ ελέγχου που θα παρακολουθούν πώ γίνονται όλα αυτά, που θα συλλέγουν στοιχεία. Μπορεί να επιχειρηματολογήσει κανεί υπέρ τη μια ή τη άλλη πλευρά, αλλά κάποιε φορέ πρέπει να δούμε τα αίτια για τα οποία διαπραγματευόμαστε και πολύ πιο σημαντικό είναι αν διαπραγματευόμαστε για του σωστού λόγου. Δεν υπάρχει πάντοτε πρόβλημα διαφθορά λόγου χάρη ή υπεξαίρεση ή κακή ε, συμπεριφορά ή παραβίαση από την πλευρά των ε, ε, αναδόχων του έργου. Τώρα, το άλλο ερώτημα που μου θέσατε είναι πολύ περίπλοκο. Γιατί μπορεί να συλλέγονται πληροφορίε και να ελέγχονται, αλλά κατά τα άλλα δεν μπορεί να δίδονται και πληροφορικά πολλέ πληροφορίε που μπορεί να ε, βοηθήσουν τι επιχειρήσει να συνεννοηθούν ε, στου διαγωνισμού. Ε, είναι πολύ λεπτή η ισορροπία και δεν ξέρω αν πρέπει να τεθεί σε επίπεδο εθνικό ή δημοτικών αρχών. Πάντω, ω τώρα δεν επιδιώκεται επαρκώ. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερε πληροφορίε σε αυτή την απάντηση. Επίση, ξεπέρασα το χρονομιλίε μου προηγουμένω. Ε, εάν είναι καλή οδηγία ή όχι η πρόταση οδηγία. Εγώ νομίζω ότι γενικά δεν είναι άσχημη. Κάποιοι ορισμοί πρέπει περισσότερο να αποσαφινιστούν. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι ευπρόσδεκτη και νομίζω ότι με λίγη δουλειά θα βελτιωθεί. Με συγχωρείτε, δεν νομίζω θα πάρω πρώτο στο λόγο, οπότε τα λέω όλα μπερδεμένα. Για τον ορισμό των εκχωρήσεων, ιδίω για το εάν εκχωρήσει πρέπει να ισχύουν για όλου του τομεί δραστηριότητε, όλε τι κοινοφιλήσει και δημόσιε υπηρεσίε, η απάντηση είναι όχι διότι υπάρχουν διαφορετικές ε, μορφές ε, εταιρικών σχέσεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και αυτό ισχύει και τις εκχωρήσεις όπου ε, ο κίνδυνος μεταφέρεται βάσει κάποιας αίτησης όμως ουσιαστικά, κάποια βάση συνεννόησης. Υπάρχουν όμως άλλες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, τα νοσοκομεία, οι φυλακές όπου υπάρχουν άλλου είδους συμβάσεις. Περιλαμβάνεται και πάλι ιδιωτικός τομέας τομέα στην παροχή της υπηρεσίας αλλά δεν εννοούμε αυτό με τις κατεκχώρησης συμβάσεις. Θα πρέπει να πλαισιωθεί όλο αυτό σε διαφορετικό τρόπο. Για τον νόμο ΣΑΠΑ ε, είπα ότι μάλλον ήταν πιο διαλεκτικό, πιο ευέλικτο από την σημερινή πρόταση οδηγία. Ω προ το κείμενο, ε, στον νόμο αυτό πραγματικά δεν υπάρχει υποχρέωση κριτηρίων ε, ένωση όταν και ανάθεση όταν γίνεται η εξέταση των προσφορών, αλλά αυτό γίνεται σχεδόν αυτομάτω. Το πεδίο εφαρμογή βέβαια δεν είναι τόσο διαφορετικό από εκείνο τη οδηγία, ό,τι αφορά τι τιμέ αναφέρθηκε αν θα πρέπει να περνάμε από τον ιδιωτικό το δημόσιο τομέα προ την διαδικασία ανάθεση. Εδώ, σε γενικέ γραμμέ, όχι ειδικά για αυτήν την οδηγία, τι συμβαίνει. Ότι στην περίπτωση τη υδροδότηση στη Γαλλία, με τι διατάξει που έχουμε, είχαμε άψογα αποτελέσματα. Διότι συχνά οι φορεί τοπική αυτοδιοίκηση αναθέτουν τι συμβάσει με πολύ συγκεκριμένε τιμέ και όχι με τυχαία ποσά. Άρα οι ιδιώτες το καθορίζουν αυτό με πιο περιπλοκές υπηρεσίες, πιο ε, δαπανηρές και με δυσκολότερο σύστημα παροχή. Άρα δεν είναι τόσο απλό να πούμε θα πρέπει να καθορίζεται από την ιδιωτικότητα ή τομέα. Ε, υπήρχαν και άλλε ερωτήσει, αλλά ήδη έχω ξεπεράσει το χρόνο ομιλία μου. Ευχαριστώ. Νομίζω, εκεί, εσείς κύριε Βαρχοβάν έχετε τις περισσότερες ερωτήσεις. Δεν είχα κάποια συγκεκριμένη ερώτηση εγώ, γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομο. Απλώ να επαναλάβω ότι οι βασικέ αλλαγέ που χρειάζονται στην πρόταση οδηγία είναι η διαδικασία ανάθεση, όπου θα έλεγα όχι, να μην περάσετε στην κατεύθυνση των δημόσιων διαγωνισμών, αλλά να είναι ποιότερο το καθεστώ. Διαφορετικό ε, τομέα είναι αυτό. Ε, υπάρχουν κάποιε κοινέ διαδικασίε βέβαια, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε κυρίω τη διαφάνεια και αυτό θα πρέπει να είναι η βασική μα μέρημνα. Δεύτερο στοιχείο καταλαβαίνω ότι για το κάθε διαφορετικό τομέα θα ισχύουν και διαφορετικά επίπεδα ε, αξία. αλλά αυτό είναι σημείο καθοριστικό. Αναφέρθηκε το θέμα τη διάρκεια. Η διάρκεια, νομίζω, σωστά έχει περιγραφεί στην Οδηγία ω Γενική Αρχή. Είναι κάτι που καλωσορίζουμε. Και τέλο, νομίζω ότι πρέπει κάποια από τα δύσκολα στοιχεία της μετατροπής ε, να βγουν από την οδηγία, διότι η επαναδιαπραγμάτευση είναι ο κανόνα στην πράξη, αντί, για να είναι, αντί εξαίρεση, όπως ο είπε ο συνάδελφος. Ευχαριστούμε. Κύριε Βέιαντ. Θα προσπαθήσω και πάλι να πάρω μια θέση για τα σημεία που αναφέρθηκαν. Ένα πρώτο σημείο είναι η συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες. Μα εδώ είναι σαφές ότι ένας Δήμος μπορεί να αποφασίσει για το θέμα αυτό, αλλά η οδηγία αυτή όμως οδηγεί ότι όταν οι Δήμοι και οι κοινότητες ε, θέλουν να εφαρμόσουν αυτήν την ε, εφαρμογή της οδηγίας, δεν έχουν καμιά δυνατότητα να επιτρέψουν μια συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αυτό λοιπόν δεν οδηγεί σε μια μεγαλύτερη ε, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, οι Δήμοι έχουν πάντα την δυνατότητα, δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την, ε, ιδιωτική συμμετοχή για να έχουν μεγαλύτερη ευκαμψία. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν ιδιωτικέ ε, συμφωνίε, παραδείγματο συμφωνίε με τον ιδιωτικό τομέα για την υδροδότηση και βάσει των, ε, της οδηγίας αυτής όταν εκπνέει αυτή η συμφωνία είναι, δεν μπορούν τίποτα να κάνουν οι δήμοι για να κρατήσουμε αυτήν την ε, σύμβαση. Και επιπλέον στη Γερμανία υπάρχει το πρόβλημα πολλών εταιριών που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ε, υδροδότησης ε, θα υπάρξει ουσιαστικά έξοδος από το κρατικό μονοπόλιο και αυτό θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα τα οποία θα υπάρξουν και στον ενεργειακό τομέα στην Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε λιγότερη συμμετοχή σε εταιρικέ σχέσει ιδιωτικού και δημόσιου τομέα από ό,τι στο παρελθόν. Και αναφέρθηκε και το θέμα του οδηγού. Για μένα η διαφορά των συνθήκων, των συμβάσεων εκχωρήσεως είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα Στη μία περίπτωση τη συμβάση, παραδείγματο χάρη προμήθεια, υπάρχει ένα στόχο, ενώ στην περίπτωση αυτών των συμβάσεων εκχώρηση υπάρχει μια συνεχή παροχή υπηρεσιών και για μένα αυτή είναι η, αυτή η αποχρούσα διαφορά αυτών των συμβάσεων από τι συμβάσει τη Η κυρία Σιμών θα ήθελε να πει κάτι. Ένα λεπτό το πολύ. Ναι, πολύ σύντομα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Σουσιέ για την ιδιαιτερότητα των εκχωρήσεων και το χρόνο που χρειάζεται για να προσαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα. Οι διατάξεις για την εκτέλεση των εκχωρήσεων που προβλέπει η πρόταση στο άρθρο 42 πρέπει να αναθεωρηθούν σοβαρά για να ανταποκρίνονται καλύτερα στην ιδιαιτερότητα αυτή. Και κάτι άλλο για τις διαφορές που υπάρχουν και ολόκληρη την γάμα των υπηρεσιών που προσφέρονται. Αυτό ακριβώς είναι επιχείρημα για την light approach που λέμε. Χωρίς να μειώνεται η διαφάνεια βέβαια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας κύριε Πρόεδρε για την ίση μεταχείριση. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχω γίνει θύμα άνησης μεταχείρισης. Η συζήτηση έδειξε ότι το θέμα είναι πολύπλοκο και αφορά πολλές και διαφορετικές καταστάσεις. Είναι δύσκολο να διευθετηθεί αφηρημένα Μόνο δύο λύσεις βλέπω. Η μία είναι αυτή που είπε ο κύριος Φερχούφεν, την light approach δηλαδή. Δεν μπορούν να καλυφθούν όλα με ένα νομοθέτημα. Δεύτερη δυνατή λύση, συγκεκριμένοι κανόνες για συγκεκριμένες καταστάσεις ή τομείς. Ευχαριστώ. Μπένετ. Ο κύριος Βαμπ ρώτησε κάτι πολύ θεμητό. Αν η επέκταση των κανόνων του δημόσιου τομέα και σε αυτές τις εκχωρήσεις θα βασίζονται ή όχι στους κανόνες των δημοσίων προμηθειών. Τυπικά ναι, αλλά το θέμα εδώ είναι υπάρχει επαρκής ευελιξία στους κανόνες δημοσίων προμηθειών για να ισχύσει και για αυτόν τον τομέα. Αν δούμε τι λέει η έννοια του ανταγωνιστικού διαλόγου, αυτή μπορεί να τα καλύπτει όλα. Μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. Τυπικά λοιπόν ναι, ναι θα επεκτείνει το δημόσιο, το πρότυπο των δημοσίων προμηθειών. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες. Ήταν εξαιρετικά όλα αυτά που ακούσαμε. Τώρα η κυρία Σικόρσκα και μετά ο κύριος Ζουβά. Παρακαλώ, σε λίγο θα ψηφίσουμε. Καλό είναι που είμαστε τόσο πολλοί να ακούσουμε τα συμπεράσματα, αλλά παρακαλώ να μην θορυβείτε τουλάχιστον. Κυρία Σικόρσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάντοτε πολύ ευχάριστο να συμμετέχει κανείς στις συνεδριάσεις σας. Ε, σας ευχαριστώ και για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης που όπου ακούσαμε τόσο διαφορετικές απόψεις. Πολλές φορές ήταν και αντιφατικές μεταξύ τους και πρέπει να πω ότι δεν μας εκπλήσει αυτό. Διότι η συζήτηση αυτή αντικατοπτρίζει αυτά που ακούσαμε τα τελευταία δύο χρόνια όσο συζητούσαμε την οδηγία αυτή. Το περιεχόμενο της και η φιλοσοφία της ε, αντικατοπτρίζουν ακριβώς τις δύσκολες επιλογές που χρειάστηκε να κάνουμε όταν επεξεργαζόμασταν το κείμενο. Ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι η οδηγία αυτή θα εγκριθεί εύκολα το αντίθετο μάλιστα. Υποβάλαμε κείμενο που κατ' εμάς αντικατοπτρίζει ακριβώς τις ανάγκες και τα θέματα που πρέπει να φυγούν. Μερικά συγκεκριμένα που είπαν οι εμπειρογνώμονες για το περιεχόμενο του κειμένου. Από τη μία λένε ότι είναι πολύ ελαφρύ το περιεχόμενο αυτό ότι πρέπει να μοιάζει περισσότερο με την οδηγία των δημοσίων προμηθειών. Από την άλλη όμως ακούγεται μια άλλη φωνή που ζητάει πολύ διαφορετικό τρόπο διευθέτησης των εκχωρήσεων και αυτή είναι νομίζω η πλειοψηφία. Νομίζω πάντως ότι όσο μεγάλη και να είναι η διαφορά αυτή θα λυθεί με περισσότερη διαφάνεια και όχι με λιγότερη. Γιατί εδώ χρειάζεται απλοποίηση, το streamlining που λένε. Για την απελευθέρωση της αγοράς δεν αρκεί ποτέ να λέμε ότι η αυτή δεν αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ούτε τη δομή συγκεκριμένων αγορών. Ένας από τους ομιλητές είπε ότι πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε τομείς όπως το νερό. Αυτό απαιτεί ακριβώς περισσότερη έρευνα γιατί δεν θα υπάρξουν τόσες επιπτώσεις όσες αναφέρθηκαν. Δεν καλύπτονται όλα από αυτή την οδηγία. Να είναι σαφές λοιπόν τι εννοούμε για τη συμμετοχή των ιδιωτών εμεί, δεν το είπε η Κομισιόν αυτά, αλλά το δικαστήριο. Κάτι ακόμη για την σαφήνεια και ασάφεια. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, όσοι θεωρούν ότι οι εκχωρήσει είναι κάτι ανάλογο με τις δημόσιες προμήθειες ζητούν αυστηρότερους κανόνες. Όσοι θεωρούν λιγότερους κανόνες θεωρούν ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Πρέπει όμως να αποφασίσουμε ποιο είναι ακριβώς το θέμα. Και από αυτό θα προκύψει η αυστηρότητα ή μη των κανόνων της οδηγίας. Τέλος, οι δύο τελευταίοι ομιλητές είπαν ότι για κάθε τομέα χρειάζονται συγκεκριμένοι κανόνες. Πρέπει να ξαναπούμε ότι η οδηγία αυτή δεν διευθετεί συγκεκριμένους τομείς είναι, αφορά αποκλειστικά τα λιμάνια, όχι κανέναν ειδικό τομέα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Σικόφσκα. Ευχαριστούμε που καθόρισατε ένα τόσο σαφές πλαίσιο. Δίκιο έχετε. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να συμβάσουμε τις διαφορετικές αυτές προτάσει. Τώρα θα ολοκληρώσει αυτόν τον γύρο ομιλίων ο κύριο Ζουδά. Σας παρακαλώ. σα παρακαλώ. Ξέρω πολύ είναι όρθιοι, Αλλά αφήστε τον εισηγητή μα να κάνει τα καταληκτικά του σχόλια. Θα ήταν ε, ευγενικό, τουλάχιστον. Κύριε Ζουβά, ευχαριστώ. Ήταν πλούσια η συζήτησή μα διότι πραγματικά είναι πολλά τα θέματα που θίξαμε. Πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσουμε την ελευθερία των δημοσίων αρχών. Ελευθερία στη διαχείριση. Ελευθερία ε, στη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό ήταν η ουσία τη συζήτηση. Δεν θέλουμε να είναι ένα κείμενο ιδιωτικοποιήσεων αυτό. Ε, δεύτερον, να εντοπίσουμε για τι ε, αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση ανά περίπτωση το τι χρειάζονται, ποιε είναι οι ανάγκε του και ποιε θα είναι οι ιδανικέ συνθήκε διαχείριση. Τρίτον, οι εκχωρήσει και αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, δεν είναι νομίζω δημόσιοι διαγωνισμοί, διότι απαιτείται εδώ ευελιξία. Χρειάζεται να είμαστε διαλεκτικοί. Και συνέπεια της ευελιξίας είναι η διαφάνεια. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι για να την πετύχουμε. Τέταρτον, οι εκχωρήσει, ακριβώ επειδή είναι συμβάσει πολύ μεγάλη διάρκεια κάποιε φορέ, 50 χρόνια για ένα αυτοκινητόδρομο πρέπει να μπορούν να ε, τύχουν επαναδιαπραγμάτευσης. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, ως βουλευτής, προτιμώ να ψηφίσω νόμο παρά να ε, τα αφήσω όλα στη διακριτική ευχαίρεια της δικαστικής αρχής, ακόμη και αν είναι συνετή αυτή. Ευχαριστώ κύριε Ζουβά. Σας ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την ακρόαση. Νομίζω ότι ήταν ε, πραγματικά μια ιδανική, ένα ιδανικό παράδειγμα για το πώς θα πρέπει να διεξάγονται οι ακροάσεις. Πολύ ωραίες και διαφορετικές απόψεις. Η κυρία Βερνιό είπε ότι περισσότερες ε, απορίες έγινε παρά έδωσε απαντήσεις. Αυτό είναι καλό και θα ήθελα τώρα να χειροκροτήσουμε τους εμπειρογνωμονές μας σήμερα. Το αξίζει. Um, and um, just, uh, we should just close, I think, Philip και απλώς, κύριε Ζουβάν, να θυμίσουμε το χρονοδιάγραμμα για την πρότασή σας. Θα μου τα δώσει εδώ η Μαγλή. Το δικό σας σχέδιο έκθεση θα αποσταλεί στις μεταφραστικές υπηρεσίες 25, στις 25 Απριλίου. Πρώτη εξέταση 29 Μαΐου 21 Ιουνίου προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ, το Σεπτέμβριο, θα συζητήσουμε τι τροπολογίε. Ανυπομονούμε λοιπόν να ξεκινήσει όλο αυτό το έργο. Είμαστε δεσμευμένοι και ευχαριστούμε και όσου μα παρακολούθησαν στο διαδίκτυο σε αυτή την ακρόαση. Τώρα θα συνεχίσουμε. Θα κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, γιατί ξέρω ότι πολλοί δεν μένουν για τι ψηφοφορίε. Κάποιοι έρχονται, οπότε θα ε, συνεχίσουμε σε πέντε λεπτά με την ψηφοφορία που θα δώσω το λόγο στην κυρία Κόμη. I don't. No, you keep that. Okay. Uh, could I invite everybody to take their places, please? Παρακαλώ να λάβετε θέσεις για να αρχίσει η σημαντικότατη αυτή ψυχοφθορία. Eleven Κυρίες και κύριοι μου, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της σημαντικότατης αυτής πρότασης από την Κομισιόν για την τυποποίηση. Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά του την ομάδα της Κομισιόν εδώ, που όπως πάντα προσέρχεται να παρατηρεί. Η συγγήτρια μας είναι η κυρία Κόμη Πρώτα όμως καλωσορίζω θερμά για πρώτη φορά από την εκλογή της τον αντιπρόεδρο, τον αντιπρόεδρό μας Πετικάινεν, την κυρία Πετικάινεν. Έχουμε και ένα νέο συνάδελφο από τη Γερμανία. Την επόμενη φορά θα την παρουσιάσω. Λοιπόν, τώρα, κυρία Κόμη θέλετε να κάνετε καμία προκαταρκτική δήλωση πριν την ψηφοφορία. Βεβαίω, ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες για τη στήριξή τους ε, κατά την επεξεργασία των τροπολογιών, των συμβιβαστικών τροπολογιών. Δυστυχώ, οι ληστές δεν προσυπέγραψαν την τροπολογία για την ε, δυνατότητα συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ελπίζω όμω θα βρούμε μια κοινή θέση προκειμένου να δώσουμε ένα σαφέ μήνυμα προ του εθνικού οργανισμού τυποποίηση, ώστε να προχωρήσουν και να κάνουμε ένα βήμα προόδου, να απλουστευτεί επιτέλου το σύστημα. Uh, any other shadow η κυρία Ρούλα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Κόμη, γιατί στο τέλος καταφέραμε να καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές λύσεις και αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες οδήγησαν να αποσυρθούν παλές τροπολογίες και ε, το έχω πράξει αυτό ήδη. Αν χρειαστεί να αποσύρουμε και άλλες θα το πράξω. Όπως είπα όμως έχω αποσύρει ορισμένες τροπολογίες. Άμα χρειαστεί θα λάβω το λόγο σχετικά. Και έχω και μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία 27. Σας ζητώ να μου δώσετε το λόγο όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Κόμη και για τη συνεργασία αυτή. Ναι, θα έχω το μυαλό μου, λέει ο κύριο Μάλκον. Κυρία Μόζερ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λάρα Κόμη και όλες τις, όλους τους κοιόδης για τη συνεργασία τους. Ξέρω ότι είχαμε κάποιες δυσκολίες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό και το υποστηρίζω. Θα ήθελα απλώς να πω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πράγματι <clears throat> μια καλύτερη πρόσβαση στα θέματα τυποποίησης, εναπόκειται φυσικά στα κράτη-μέλη και τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, να δουν το πώς θα το πετύχουν αυτό και αν έχουν χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής θα πρέπει να πάρουν τις απαραίτητες αποφάσεις. Γενικά όμως υποστηρίζουμε την λύση και την έκθεση κόμι γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Κόμη για το πνεύμα ε, συνεργασίας που μας οδήγησε στην τελική συμβαστική λύση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος Μάλκομ Χάρμπορ. Ναι και οι άλλοι σκιώδεις. Και ελπίζω οι κόρη σας να είναι καλύτερα γιατί χρειάστηκε να φύγετε. Χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι. Ναι, είχε ε, έκανε μια εγχείρηση χθε το βράδυ. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Λάρα. Και και τους κοιόδης εισηγητές. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ήταν ευτυχές. Κάποιες στιγμές εγώ διαμαρτυρήθηκα ότι ίσως κάνουμε πολύ πολύπλοκη την νομοθεσία και ως νομομαθής πιστεύω ότι πρέπει να είναι λειτουργική η νομοθεσία, στην πολιτική δεν είναι πάντα εύκολο να το πετύχει κανείς αυτό. Νομίζω τελικά ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι με το τελικό αποτέλεσμα. Και ο Έντουαρτ, ο οποίος ήταν εισηγητής για την ειδική έκθεση. Ε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, να τονίσω απλώς ότι οι κύριες αρχές της έκθεσής μας έχουν εξασφαλιστεί Φτάνουμε στο τέλος αυτού του έργου που χρειάστηκε σχεδόν τρία χρόνια και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την Επιτροπή μας γιατί αυτό είναι ένα νέο νομοθέτημα μετά από πολλά χρόνια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία. Και εγώ θα είμαι ο τρίτος ψηφοφόρος της ομάδας μου. Άρθρο ένα παράγωγος ένα από ό,τι καταλαβαίνω η κυρία Ρούλα έχει αποσύρει την τροπολογία της 111. Πάμε στην 112 στην περίπτωση αυτή. ψήφι υπέρ. Α, και αυτή για αποσυρθεί. Ωραία. Τι να κάνουμε, εγώ φταίω. Βιομηχανία 20. Ψήφι υπέρ. Α, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά για την 20 ε, της βιομηχανίας. Πέρα τη ψηφοφορία. 25-17 κατά γίνεται δεκτή. Και στη συνέχεια πάμε στο άρθρο 2. 119. Ζουβέν και Κόμι. Υπέρ, κατά, αχές, δεκτή. Εκπίπτουν οι δύο τροπολογίες που ακολουθούν. Τροπολογία 121 Κοχμερίν σαν προσθήκη ψηφίπερ Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. 121 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Ε. Ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. 1-2-2, Σαλβίνι, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται σαφώς. 123, Ρούλε Τούρνεν. Άρχεται για 123. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 κατά δεκτή. Συγγνώμη, συγγνώμη, έχασα τις πίσω μου σελίδες. 124 της κυρίας Άνσλικ. Γιατί 123 δεν είναι κρίτη. 124 Χάνσλικ. Ψήφι υπέρ. Ηλεκτρικά. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίβεται. 19 ακόμη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Α, δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 21 και 22 Ήτρε. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 128 Σαλβίνη σαν προστίκη υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 22 κόμι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 129 Ρούλε και άλλων σαν προστίκη άρχεται ηλεκτρονικά πέρας Απορρίπτεται. 23 οι κόμοι και οι ε, άλλες υπέρ κατά δεκτή. 1.31 Σαρντεμόζε. Ηλεκτρονικά αρχίζουμε για την 131. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 κόμοι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 132 και 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεκτές 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οι 136-135 έχουν αποσυρθεί. 137 Σαντεμόζε άρχεται. Ηλεκτρονικά. πέρα στι ε, ψηφοφορίε, απορρίπτεται. 26 κόμι υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 138 Σαλβίνη υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 139 Δε άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 139. Πέρας απορρίπτεται. 24 Ήτρε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ίσως ο συντονιστής του έρθει να μας δίνει σήμα λίγο νωρίτερα. Απορρίπτεται. 25 Ήτρε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. απορρίπτεται. Βιομηχανία 26 ηλεκτρονικά υπέρ κατά απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 141 Ροσφόρ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 με το προφορική τροποποίηση της κυρίας Ρούλα. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, καλά. 27 εκπίπτει. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1.47 Σαλντεμόζε υπέρ κατά αποχές δεκτή εκπίπτει 28, 29 βιομηχανία υπέρ κατά δεκτή. Έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος. Α, ήσασταν κατά, δεν σας κατάλαβα. 29 βιομηχανία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασμα. Απόλυτα. Διεθνές εμπόριο 12, σαν προσθήκη. Υπέρ. Εντάξει, την ψηφίζουμε. Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι. 148 Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. 149 και 150 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 29 και 28 εκπίπτουν. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 181. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα 181. Πέρας. Απορρίπτεται. Βιομηχανία 30. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε στην 163. Αποσύρεται. 160. De Jong. Άρχεται η ψηφοφορία για τα 160. Πέρας. Απορρίπτεται. 161. De Jong. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 162. Κροσφόρ. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 20-17. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 100. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 165. De Jong. Άρχεται. Πέρας απορρίπτεται. 164 ρούλα και του όρων, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 166 De Jong, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14, υπέρ, Α, να ελέγξουμε, εντάξει. Συμβαστική 14, έλεγ, ε, άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 34 ακόμη, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Εκπίπτει 15 ΣΥΝΤΑ, τροπολογία 35 της εισηγήτριας, υπέρ, Έχετε αποσύρει, εντάξει. Ε, 182-183 είναι ταυτόσιμες, ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ίντα 16 υπέρ. Όχι, ψηφίζουμε και εδώ πάλι ηλεκτρονικά. Είναι τα 16, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 37 κόμι, υπέρ. Κατά. Δεκτή. Εκπίπτει είναι τα 18, είναι τα 17. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 38 κόμι, υπέρ. Κατά δεκτή συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 191 ναι 191 Ζουβέν υπέρ κατά αποχές δεκτή 195 Ρούλα υπέρ. Μάλλον άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ήτρε 37. Άρχεται η ψηφοφορία για την Ήτρε 37. Πέρασε. Απορρίπτεται. 196 Σαλτεμόσε και Ήτρε 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 197 και οι υπόλοιπε εκπίπτουν. Συμβιβαστική τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 202 Σαλτεμόσε υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 203 έχει αποσυρθεί από τους πράσινους. 2-4 Ζουβέν υπέρ κατά αποχές δεχτεί. Εκπίπτει η Ήτρε 39, 205 έχει αποσυρθεί, 206 Ζουβέν υπέρ κατά αποχές δεχτεί. 40 εκπίπτει, 207 κόμι υπέρ κατά αποχές δεχτεί. 41 του συζήτρια υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά δεκτή. Πάμε στη 212. Έπεσε ή στέκεται. 212. Άρχεται η ψηφοφορία για την 212. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. Εγώ την υπέβαλα, αλλά δυστυχώς πρέπει να την απορρίψω. 42 από τον εισηγητή. Διεθνές εμπόριο. 42. άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτονται 208 ρούλα και οι υπόλοιποι άρχεται η ψηφοφορία ρούλα και λοιποί. πέρας εγκρίνονται Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. 20 υπέρ κατά εγκρίνεται 2 21 Μάντερ υπέρ κατά απορρίπτεται 222 νομίζω για να πέσει η κυρία Σαδεμόζε 21 συμβαστική 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 συμβαστική 22 υπέρ κατά εγκρίνεται 230 πάει και λοιπή. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Είναι 25 ως προσθήκη. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 23. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και τώρα 235 Σαλβίνη υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 46 της εισηγήτριας υπέρ, άρχεται μάλλον η ψηφοφορία για την ε, 46 πέρας εγκρίνεται 236 το κύριο Ροσφόρ υπέρ κατά εγκρίνεται 47 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται 48 της εισηγήτριας υπέρ άρχεται μάλλον η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 237 υπέρ κατά απορρίπτεται. 238 πάξα υπέρ κατά εγκρίνεται. 239 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά εγκρίνεται. 242 πάξα, υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά εγκρίνεται. Επιτροπή Βιομηχανία 46 υπέρ. Νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 46 τη βιομηχανία, υπέρ. Συγγνώμη, πέρας. Απορρίπτεται. 47. Διαγραφή που προτείνεται από τη βιομηχανία υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 50 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 51 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 246 της εισηγήτριας. Άρχεται η ψηφοφορία για την 246. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 52 τη εισηγήτρια. Επιτροπή Βιομηχανία 48. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Διεθνέ εμπόριο 27 ω προστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Διεθνέ εμπόριο 28. Υπέρ. Άρχεται μάλλον η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 247 αποσύρεται. 248 σαλτεμόζε υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 53 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 54 εισηγήτρια υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 49 ήτρε εκπίπτει. 55 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 50 ως προσθήκη Άρχεται η ψηφοφορία. Ήτρε 50 ως εκεί. Πέρα. Εγκρίνεται. 56 εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 249 σάλτεμο της εισηγήτριας. Συγγνώμη της κυρίας Σαλντεμόζε. Σκέω της εισηγήτρια τέλο πάντων. Λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με διαφορά. Ήτρε 51 εκπίπτει, 57 της εξηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 251 της κυρίας Άλντεμόζε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 251. Πέρας. Απορρίπτεται. Βιομηχανία 52 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 58 της εισηγήτριας. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 58 της εισηγήτριας, πέρας. Εγκρίνεται. 59 της εισηγήτριας, υπέρ. Άρχεται μάλλον η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 60 της εισηγήτριας, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 252 Εκπίπτει 253 Σαλβίνη. Υπέρ. Κατά. απορρίπτω την αδιάφορα. 255 εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 61 και 254 εκπίπτουν. 62 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 256. Ζουβα, Άρχεται η ψηφοφορία για την 256. Πέρας. Απορρίπτεται. 63 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 64 και 257 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Διεθνέ εμπόριο 30 κρύπτει. 31 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Βιομηχανία 54 υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε. Υπάρχει πρόβλημα. Ηλεκτρονικά. Ήτρε 55. Ήτρε 55. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 251. 59 δεγιόν. Άρχεται η ψηφοφορία για το 259. Πέρας. Απορρίπτεται. 260 της κυρία Ζούλα και της κυρία Τουρούναν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται με διαφορά. Διεθνές εμπόριο 32. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 262 του κυρίου Ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 261. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 263 υπέρ κατά απορρίπτεται. 264 υπέρ κατά εγκρίνεται. 265 ως προστίκη. Άρχεται η ψηφοφορία. 265. Πέρας. Εγκρίνεται ως προστίκη. Ήτρε 56. Ως προστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 65. Της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 266. Το κύριο Ροσφόρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά εγκρίνεται. 2,69 και 2,70 υπέρ κατά εγκρίνονται. 2,72 υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 272. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. So they all fall. Sorry. Yeah. All right. Okay. All right. Okay. We'll close the vote. And that's rejected. Απορρίπτεται. Με συγχωρείτε, είχαμε κάτι διαβουλεύσει. Απορρίφθηκαν τέλος πάντων. 275. And we need to All right. Okay. Sorry, we, we just need to uh, just clarify that. We rejected 272. Η 272 απορρίφθηκε. Όμως θα ψηφίσουμε τις υπόλοιπες. Η 271 λοιπόν. Σαλντεμόζε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 271. Πέρασε. Απορρίπτεται. 273. Το κύριο Κουπάκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται επίσης. 274 της κυρίας Ράπτη. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πρέπει να τις ψηφίσουμε όλες. Πέρας. Απορρίπτεται και αυτή. Όλες οι τροπολογίες απορρίφθηκαν για το παράρτημα 3 σημείο D2. 275. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 276. Με ένα τεσχυρόν υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται με διαφορά. Αιτιολογικές σκέψεις. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 70 σαλτεμόζε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ήτρε 3 επίπτη. Ίντα 2. Άρχεται η ψηφοφορία για την Ίντα 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Είναι τα τρία. Υπέρ. Όχι να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία για την είναι τα τρία. πέρας. Εγκρίνεται. Είναι τα τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Να, επιταχύνουμε λίγο. Ας ψηφίσουμε για την 94 ηλεκτρονικά. Uh, the vote is closed. Έληξε. Εγκρίνεται 19-16. Τώρα 71 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 74. Ηλεκτρονικά. άρχισε, έληξε, απορρίπτεται. Ξανά ηλεκτρονικά 75. 75 έληξε απορρίπτεται ηλεκτρονικά 76 α όχι ηλεκτρονικά κατά κατά είπα Απορρίπτεται. Εβδομήντα οχτώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. Βιομηχανική 4. Ηλεκτρονικά. έληξε απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται 81 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται βιομηχανική 5 συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 87 και 88 ταυτόσημα. άρχεται η ψηφοφορία έληξε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 101 άρχεται έληξε απορρίπτεται Έξι υπέρ κατά εγκρίνεται 104 άρχεται η ψηφοφορία έληξε απορρίπτεται 105 άρχεται η ψηφοφορία έληξε Απορρίψατε. 106 λοιπά. Άρχεται. Τον 6 είπα και 10. Έληξε. Α, εγκρίνεται πανηγυρικά. 7 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται 8 υπέρ κατά εγκρίνεται 11 της βιομηχανίας ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται 9 υπέρ κατά εγκρίνεται 10 υπέρ κατά εγκρίνεται 107 υπέρ κατά εγκρίνεται 11 και 12 υπέρ κατά εγκρίνονται επτά κατά πίπτη δώδεκα υπέρ κατά εγκρίνεται βιομηχανική δεκατέσσερα ηλεκτρονικά έλεξε εγκρίνεται με δύο ψήφους πλειοψηφία δεκατρία υπέρ τα εγκρίνεται βιομηχανική 16 υπέρ κατά εγκρίνεται 108 βιομηχανική 16 άρχεται η ψηφοφορία έληξε εγκρίνεται 108 άρχεται. Έληξε, απορρίπτεται. δεκατέσσερα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. δεκαπέντε υπέρ, κατά, εγκρίνεται δεκαέξι. α. Θέλετε ξανά τη 15, καλά τη 15 ξανά ηλεκτρονικά. Έλξε. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Βιομηχανική 18 υπέρ κατά εγκρίνεται. Μα συνεχώς αλλάζεται βλέπω. Βιομηχανική 18 ηλεκτρονικά. Έλξε. Εγκρίνεται. Άρα η 109 καταπίπτει. Καταπίπτει. 110 υπέρ. Όχι, άρχεται η ψηφοφορία. Για την 110. Ψηφίζετε όλοι. Άρχεται η ψηφοφορία 110. Έληξε. Μάλιστα, εγκρίνεται. Δεν ψηφίσαμε την 109. Λέει καταπίπτει αν η ίδια εγκρίνεται. Χαίρομαι που διαβάζετε με τέτοια προσοχή. Εννοεί αν είχε εγκριθεί η βιομηχανική 18. Τι, να, τι λέει η κυρία Ρούλα. Για την 109 λέγαμε και η ακόμη εννοούσε την 18 ρε παιδιά. Ευχαριστώ όμως τον συντονιστή για την προσοχή του. 10 ψηφίσαμε, εγκρίναμε, μάλιστα. Μάλιστα. Ποιος ήθελε να την αποσύρει. Θέλετε να το ξανακάνουμε, να ξαναψηφίσουμε. είχε εγκριθεί 110. Βιομηχανική 19 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τελευταία τροπολογία η 17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα. Τώρα λέγω το σύνολο. Το σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία για το σύνολο έληξε εγκρίνεται 36 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια. Παρακαλώ ησυχία. Εισηγήτρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες και τις πάσες για τη συνεργασία μας γιατί εγκρίθηκαν τόσο πολλοί συμβιβασμοί. Είχα προτείνει και εγώ να εγκρίνουμε ήδη από την πρώτη ανάγνωση για να επιταχυνθεί λιγάκι η διαδικασία της έγκρισης. Προτείνετε λοιπόν, θέλετε εντολή για να δούμε τι φρονούν οι πολιτικές ομάδες γιατί οι συντονιστέ πρέπει να τα αποφασίσουν αυτά. Κυρία Γκέπχαρτ ή κυρία Σαλντεμόζερ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κόμη για την πολύ καλή συνεργασία και χαιρόμαστε γιατί καταφέραμε χθες έστω και την τελευταία στιγμή να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις που μπορούν να υποστηριχθούν από όλους. Βέβαια είναι πολύπλοκο το κείμενο και η ομάδα μου θα ήθελε να ελέγξει λιγάκι το κείμενο όπως έχει προκύψει από την ψηφοφορία να δούμε γιατί έχουμε κερδίσει κάποιες τροπολογίες, έχουμε χάσει κάποιες άλλες τροπολογίες. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να αναλύσουμε καλύτερα το τελικό αποτέλεσμα και γι' αυτό η ομάδα μου δεν είναι έτοιμη σήμερα να δώσει την ταχεία οδό για την, ε, για την πέραπτωση διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση και παρακαλούμε την κυρία Κόμη να δείξει λίγη υπομονή. Δεν ήταν εύκολο λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα κείμενο. Τώρα έχουμε χρειαστεί να ψηφίσουμε ένα αμφιλεγόμενο κείμενο που με δυσκολία βρέθηκαν κάποιες ε, ε τροπολογίες. Γι' αυτό δεν θέλουμε σήμερα να πάρθει απόφαση για εντολή στην εισηγήτρια για συμφωνία πρώτης ανάγνωσης. Θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Εγώ βλέπω η πρότασή μου τώρα ως εισηγητή ότι η εισηγήτρια μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ε, άτυπες αλλά τεχνικού χαρακτήρα συζητήσεις με την ε, Προεδρία για να δούμε πόσο κοντά είναι η θέση μας με τη θέση του Συμβουλίου που είναι το βασικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις για λήξη της διαδικασίας σε πρώτη ανάγνωση και η κυρία Κόμη να έρθει τότε στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών που θα είναι στις αρχές Απριλίου για να γνωρίζει κατά πόσο και αυτοί οι σκιώδεις συζητητέ μπορούν να ξεκινήσουν τι διαπραγματεύσει. Νομίζω ότι αυτό ζητάει και η κυρία Γκέπχαρτ, γιατί έτσι θα, έχουμε, θα έχουν οι πολιτικέ ομάδε το χρόνο να εξετάσουν το κείμενο. Αν συμφωνήσουν και οι άλλε ομάδε. θα πρότεινα λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία ότι η κυρία Κόμη θα έρθει στη συνεδρίαση των συντονιστών, θα προσκληθεί να έρθει και ενδιαμέσω θα πρέπει να ξεκινήσουμε τεχνικέ συζητήσει με του συντονιστέ Κυρία Μόζερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς συμφωνούμε να συμμετάσχουμε στην προετοιμασία και τις άτυπες συναντήσεις μέχρι να το συζητήσουν οι συντονιστές και συντονίστριες. Σβάμπ. Και εμείς δεχόμαστε αυτή την πρόταση. Θα ήθελα όμως η εισηγήτρια και οι σκιώδεις να συζητήσουν τις συζητήσεις ακόμα και τις τεχνικές για να μην χάνουμε χρόνο γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ευχαριστώ. Άνερς. Ναι και εμείς συμφωνούμε και δεχόμαστε την πρόταση της Λάρας γιατί πετύχαμε τόσο πολλούς συμβιβασμούς, είναι σαφής η θέση, στο μόνο στο οποίο διαφωνούμε, τα θέματα επί των οποίων διαφωνούμε τα ξέρουμε και αυτά, αλλά εσείς πάντα λέτε να αρχίσουμε με άτυπες, άτυπες συναντήσεις, τέλος πάντων, ας το δεχτούμε. Πάντα είναι χαρά η παρουσία της Λάρας στους συντονιστές. Και εμείς θα συμφωνούσαμε για την πρώτη αναγνώση και την fast track. Αλλά Παρά το ότι χάσαμε ό,τι αφορούσε τα θέματα προστασίας δεδομένων, συμφωνούμε για έγκριση με την πρώτη ανάγνωση. Και εγώ συμφωνώ, Πρόεδρε. Ωραία. Τότε πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν προκαταρκτικές συνεννοήσεις με το Συμβούλιο ούτως ή άλλως για να δούμε πόσο κοντά βρισκόμαστε. Θα χάναμε χρόνο αν τα κάναμε πιο τυπικά και επίσημα. Λοιπόν, αυτά είχαμε αποφασίσει ως διαδικασία στην Επιτροπή μας. Θα έρθει λοιπόν η Λάρα στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών σας. Υπενθυμίζω όμως ότι το κριτήριο είναι οι συντονιστές πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά πόσο κοντά είναι οι θέσεις μας με του Συμβουλίου. Τονίζω λοιπόν ότι όπως είπε και η κυρία Ρούλα, Εμείς δεχόμαστε τις εγκρίσεις και από πρώτη ανάγνωση, αντίθετα με αυτά που φρονούν συνήθως οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων που ευνοούν τη δεύτερη. Έχουμε λοιπόν σαφή εντολή να στηρίξουμε τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αφού ομόφωνα συμφώνησαν οι πολιτικές ομάδες. Είναι σαφές ότι έχουμε λοιπόν σαφή εντολή από όλες τις ομάδες. Να μην το παρεξηγήσει κανείς. Η κυρία Λάρα. Συνοπτικά, την έκκληση αυτή την έκανα γιατί από την ψηφοφορία και μετά προέκυψαν κάποιες μικρές αλλαγές. Όχι βέβαια στο γενικότερο πλαίσιο. Πέραν αυτού, να προχωρήσουμε με τις άτυπες συναντήσεις ώστε να επιταχυνθεί η πρώτη ανάγνωση. Συμφωνώ με την κυρία Ρούλε. Ναι, εδώ υπάρχουν υψηλές προσδοκίες στις διαπραγματεύσεις. Συμφωνώ μαζί σας ότι στην πρώτη ανάγνωση θα έχουμε μεγαλύτερη επιρροή. Όμως ο δημοκρατικός έλεγχος είναι πιο περιορισμένος. Λίγοι άνθρωποι παρίζονται στις διαπραγματεύσεις. Άρα διαφωνώ με τις τελευταίες σας παρατηρήσεις. Εφόσον τη θέσετε να επεξεργαστεί και η Επιτροπή, πριν να ληφθεί τελική απόφαση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας προχωρήσουμε, γιατί η κυρία Μπαστό περιμένει εδώ και πολλή ώρα για μια σημαντική έκθεση. Όσοι δεν θα μείνουν, παρακαλώ να φύγουν αμέσως. Partly, και ησύχω. Because um, I want to open a discussion. Uh, so please, um, those that are here to observe the vote, I want to give Mrs. Bastos the floor, but I'll just wait until Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Μπαστό, αλλά θα περιμένω να φύγουν όσοι ήρθαν για τι πληροφορίε. please, if you're, leaving, you please do so quietly? So, um, Παρακαλώ, φύγετε ήσυχα για να συνεχίσουμε. Um, Κυρία Μπαστός, θέλουμε να δούμε το σχέδιο έκθεσής σας. Ελπίζω ότι θα έχουμε ένα σύντομο γύρο παρεμβάσεων. Μου και ή το θέμα το ξαναδούμε και σε κατοπινό στάδιο. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για να παρουσιάσετε τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, εφόσον διεξοδικότερη συζήτηση θα γίνει σε κατοπινό στάδιο. Πιστεύω ότι θα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Το σχέδιο έκθεσης λαμβάνει υπόψη ένα θέμα ζωτικής σημασίας σε αυτή την ε, φάση της κρίσης και για τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και θέλει να δώσει κάποια απάντηση στις 20 σημαντικότερε ανησυχίε για την ενιαία αγορά. Αυτέ τις απαρίθμησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανησυχίε όχι μόνο των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δυστυχώ έχουν περάσει τουλάχιστον 20 χρόνια μετά τη δημιουργία τη ενιαία αγορά και τελικά υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ των προσδοκιών που είχαν οι πολίτες και το πώς λειτουργεί εν τέλει η ενιαία αγορά. Υπό αυτήν την προοπτική, η συγκεκριμένη έκθεση προσεγγίζει τις 20 σημαντικότερες ανησυχίες προκειμένου να θέσει το ζήτημα των τριών κενών που εντοπίστηκαν στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κενό πληροφόρησης σε σχέση με τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα από την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το, κενό της μεταφοράς και ελέγχου υλοποίησης της νομοθεσίας, της κοινοτικής νομοθεσίας από την πλευρά των κατώμελών και ένα τρίτο κενό, κενό στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές δεν εκπληρώνονται οι αρμοδιότητες που θα προσδοκούσαν τα κατημέλη και οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει πέρας. Το έγγραφο αυτό, στο οποίο βασίσαμε και το σχέδιο έκθεσης, εντοπίζει ζητήματα κλασικά από την καθημερινή λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των καθημερινών των πολιτών, αλλά και πιο ουσιώδη ζητήματα από, αυτό το, από αυτή την καθημερινότητα. Συνοπτικά, η αναγνώριση των προσόντων, η κινητικότητα των ατόμων, η επιστροφή των δαπανών υγεία, η, η ψηφιακή αγορά της Ευρώπης και η λειτουργία της, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, η ε, αγορά της ενέργειας και η φορολογία. Αυτά τα ζητήματα αναφέρονται στο συγκεκριμένο έγγραφο και εδώ αναζητούμε κάποια ε, απάντηση, κάποιες απαντήσεις. Το σχέδιο έκθεσης ακριβώς επιδιώκει να δώσει ένα σαφές μήνυμα στα κράτη-μέλη ως προς την ε, ε, ευκυβερνησία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας και να είναι πιο προσεκτικά για το πώς ακριβώς υλοποιείται. Όλα αυτά από αυτά θα εξαρτηθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οποία σε αυτή τη φάση θα μας δώσει περισσότερη οικονομική ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας. Ακριβώς σε αυτό το πνεύμα η εσωτερική αγορά θα πρέπει να λειτουργεί με τρόπο πιο ε, ομαλό, με τρόπο πληρέστερο. και να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα αυτό και τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό το σκοπό και πέραν των εισαγωγικών σχολείων και όσων αναφέρονται στην ε, έκθεση, στην αιτιολογική έκθεση, υπάρχει και ένα κεφάλαιο που αναφέρεται ακριβώς στην ε, ευκυβερνησία. Εδώ παροτρύνονται τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να υπάρξει ε, ουσιαστική μεταφορά της νομοθεσίας και να ανταποκριθούμε στην ανάγκη να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για να λειτουργεί σωστά η ενιαία εσωτερική αγορά. Για το σκοπό αυτό η έκθεση είναι συνεκτική και αναζητά απαντήσεις όχι διεξοδικές αλλά όσο το δυνατόν σφαιρικότερες σε αυτές τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί. Ευτής εξ αρχής προσπαθήσαμε να ορίσουμε τις αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σε σχέση με τις υπόλοιπες επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν. ανάλογα με τις διάφορες ανησυχίες. Έχουμε επτά ε, γνωμοδοτήσεις από κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες τελικώς θα ενταχθούν στο τελικό κείμενο της έκθεσης. Ο πρόεδρος, ο κ. Χάμπορς, ε, συνέταξε ε, επιστολή προς τους πρόεδρους των επιτροπών, ώστε να φροντίσουμε να υπάρξει συνεκτική εδώ προσέγγιση εφόσον ε, υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα ώστε να υπάρξει απαρίθμηση σημείο προς σημείο, λύση προς λύση για τις ανησυχίες που έχουν ε, συμπεριληφθεί σε αυτό το έγγραφο. Δεν θα είναι απλή η όλη διαδικασία, όμως είναι κάτι που μας προκαλεί ενθουσιασμό και έχει και συμβολικό χαρακτήρα, διότι το μήνυμα που θα προκύψει από την έκθεση αυτή θα είναι σημαντικό. Γι' αυτό περιμένω τις απόψεις των συναδέλφων για το σχέδιο έκθεσης που είναι ενδεικτικό ως προς τις κανονιστικούς περιορισμούς που ισχύουν για τον αριθμό σελίδων. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Υπάρχουν ζητήματα, σημεία, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να τα συμπεριλάβω στην αρχή. Όμως με τι τροπολογίε θα μπορούσε να γίνει η απαραίτητη προσαρμογή του κειμένου. Ποτέ δεν θα πρέπει να χάσουμε τον στόχο που θα ήθελα να συνοψίσω για να ολοκληρώσω τη σύντομη παρέμβασή μου. Να ανταποκριθούμε ταυτόχρονα και να καλύψουμε ταυτόχρονα τα τρία κενά στη λειτουργία της εσωτερικής αγορά, τα οποία είναι με σαφήνεια εντοπισμένα. Ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε Εάν δεν άρουμε αυτά τα τρία σημαντικά εμπόδια, τους τρεις φραγμούς που οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν εντοπίσει, ε, δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς. Έτσι θα χάσουμε και μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσει κάποια οικονομική ανάπτυξη η Ευρώπη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Συνοπτικά αυτό είναι το κύριο μήνυμα. Έκθεση συνεκτική, που να δώσει προσανατολισμούς, συστάσεις, ώστε ταυτόχρονα τα τρία κενά που έχουν εντοπιστεί να καλυφθούν. Σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαστός. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο το έργο σας, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν πολλές ε, γνωμοδοτήσεις στο σημείο αυτό. Θα ήταν χρήσιμο να μπορέσουν να τα δουν όλα αυτά οι σκιώδεις εισηγητές. Μπορούμε να βασιστούμε λοιπόν σε αυτά για την τελική έκθεση και φυσικά θα είναι σημαντικές οι συμβουλές. Ένα γρήγορο γύρο λοιπόν συζήτησης. Έχουμε μονάχα 12 λεπτά δυστυχώς. Ο κύριος Ρέπο είναι εδώ, ο κύριος Μάντες θα μιλήσει για τον κύριο Ρόσφο. Κύριε Ρέπο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ένα σημαντικό θέμα αυτής της έκθεσης που είναι σημαντικό το θέμα λοιπόν αυτό και ενδιαφέρει και την ομάδα μου και εμένα προσωπικά. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος εκπροσωπώ τους συντονιστές. Ο στόχος τώρα του κειμένου είναι να εξασφαλίσουμε για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις ότι θα μπορούν να απολαμβάνουν τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς. Για να επιτύχει αυτό το εγχείρημα πρέπει να εστιάσουμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, στα συγκεκριμένα μάλλον θέματα και στις, ε, στις συγκεκριμένες λύσεις οι οποίες διευκολύνουν τα πράγματα σε καθημερινό επίπεδο. Για όλες αυτές τις λεπτομέρειες λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε στα στοιχεία τα οποία βοηθούν τους καταναλωτές και δίνουν την μεγαλύτερη δυνατή ευμάρεια σε αυτούς και στην αγορά. Μπορούμε να μιλήσουμε παραγωγός χάρη για τα συστήματα επίλυσης διαφορών, τα οποία πρέπει να έχουν εθελοντικό φυσικά χαρακτήρα. Είχαμε 200.000 αιτήσει που λάβαμε στην αρχή προστασίας των καταναλωτών Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Επίσης ένα δεύτερο θέμα είναι το θέμα της κινητικότητας των Ευρωπαίων, οι οποίοι μετακινούνται για λόγους εργασίας, για λόγους ε, σπουδών και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα. Αν κάποιος αρρωστήσει, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπου και να βρίσκεται στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη σε εμά και στην ενιαία αγορά και στις δυνατότητες οι οποίες ε, προσφέρονται από αυτή την αγορά. Πρέπει ο πολίτης λοιπόν να κατανοήσει και να έχει εμπιστοσύνη σε εμάς και υπάρχουν και οι ευθύνε οι οποίες συνδέονται με την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς. Η αγορά αυτή θα πρέπει να είναι μια λειτουργική αγορά. Αλλιώς θα καταλήξουμε να έχουμε μια κατακαιρματισμένη αγορά που είναι ουσιαστικά 27 εθνικές αγορές. Θα πρέπει λοιπόν όλοι από κοινού να εργαστούμε για να προωθήσουμε τα κατάλληλα μέτρα τα οποία οδηγούν σε πρόοδο της κατάστασης του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εμά εναπόκειται να λάβουμε τις αποφάσεις που επιβάλλονται, ώστε ο καταναλωτής να έχει την ελευθερία που χρειάζεται μέσα σε μια λειτουργική εσωτερική αγορά. Χρειαζόμαστε επίσης να έχουμε και ευρύτερους ορίζοντες και εδώ υπογραμμίζω και τη σημασία του ευρώ του κοινού μας νομίσματος. Σας κατευχαριστώ κύριος Μάντερς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκπροσωπώ τον κύριο Ροσφόρ που χρειάστηκε να λείψει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση της Κομισιόν. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν οι λαοί. Άκουσα από τον Ρομπέρο ότι περίπου 50% των Γάλλων χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην Ευρώπη. Μεγάλο ποσοστό. Καλό είναι να τονίσουμε ιδιαίτερα τα τρία κύρια σημεία. Την έλλειψη πληροφοριών, το μονομοθετικό έλλειμμα Ask ourselves why it's not working. και πρέπει να ξέρουμε γιατί υπάρχουν αυτά τα έλλειμματα, τα χάσματα. Μεταξύ των συστάσεων υποστηρίζουμε την ολιστική προσέγγιση της ενιαίας αγοράς, ότι το σημαντικότερο είναι η λαοί, γιατί χωρίς καταναλωτές και καταναλώτριες δεν υπάρχει οικονομία. Απλοποίηση επίσης της νομοθεσίας είναι απαραίτητη. Στόχος καλύτερη συνεργασία και βέβαια η ενδυνάμωση και δημοσιοποίηση των εργασιών του Λίστο, Solvit. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε την εφαρμογή των νομοθετημάτων που αφορούν την ενιαία αγορά. Έχω μερικές απορίες είδα στο σημείο 27 ότι η συγκητή ζητάει νέα πράξη για την ενιαία αγορά, αλλά αφού ακόμα ισχύει η προηγούμενη, γιατί χρειάζεται και νέα, δεν τελείωσε. Εμείς θέλουμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν και νέες πληροφορίες, ε, καμπάνιες πληροφόρησης για να εξηγήσουν στον κόσμο πόσο σημαντική είναι η ενιαία αγορά, πόσο ωραία είναι η εσωτερική αγορά. Γιατί ο κόσμος δεν αισθάνεται, δεν, βλέπει, δεν το βλέπει να δουλεύει, δεν βλέπει να δουλεύει. Χρειάζονται λοιπόν καμπάνιες για να μπορεί ο κόσμος να είναι πιο περήφανος για την Ευρώπη του. Αυτά ήθελα να σας πω. Αλλά υποστηρίζω τον εισηγητή. Η κυρία Ρούλα. Θα είμαι συντομότατη. Έχω κάποια προβλήματα με την έννοια του κενού νομοθεσίας ή του χάσματος νομοθεσίας. Αυτό είναι κάπως ε, μονομερές. Γιατί πρέπει να δούμε τα πράγματα με προοπτική και ισορροπία. Οι πολίτες φοβούνται εξίσου το κενό νομοθεσία και την υπερβολική νομοθεσία. Όπως είδαμε και με τις ακροασει προηγουμένω για την πρόταση τη Κομισιόν, η οποία ζητά να υπάρξει μια κεντρική ρυθμιστική αρχή. Υπάρχουν αμφιβολίε. Θα πρέπει να ελέγξουμε αν τα νομοθετήματα τα οποία προτείνονται, αν είναι λυσιτελή, αν πράγματι διατηρούν και τα δικαιώματα αυτοδιοίκησης των τοπικών αρχών αυτοδιοίκησης. Δεν νομίζω ότι μπορούν όλα να λυθούν τα προβλήματα με καλύτερο τρόπο στην Ευρώπη. Πρέπει να μπορεί να παραμείνει η δυνατότητα να λύνονται με καλύτερο τρόπο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εγώ θα ήμουν ιδιαίτερα προσεκτικό με την έννοια αυτή του χάσματο νομοθεσία, γιατί η υπερβολική νομοθεσία δεν φαίνει την Ευρώπη κοντύτερα στου πολίτε, αλλά μακρύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δε Γιόγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Συμφωνώ. Το Συμβούλιο, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να έχουν καλύτερη ποιότητα νομοθεσίας. Τώρα, για τις εξαρτίες συνειδητοποίησης και ε, διαφωτισμού. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες θέλουν να τους πληροφορούμε απλώς. Θέλουν να ακούγεται η γνώμη τους. Και εδώ είναι το σημαντικό στοιχείο, είναι η διάδραση με τους πολίτες, η αλληλεπίδραση. Όχι απλώς να στέλνετε ένα μήνυμα από τις Βρυξέλλες στους πολίτες και έκανα κάποιες τροπολογίες σχετικά. Τρίτο σημείο. Αν θέλουμε να ακούσουμε τους πολίτες, ένα από τα θέματα που τους ενδιαφέρουν είναι η κινητικότητα η προβληματική παραγωγή του Μόντι 2. Υπάρχει το θέμα της ε, εκμετάλλευσης των εργαζομένων, η ψευτο αυτοαπασχολούμενη, η προσωρινή εργασία, η αποσπάσεις εργαζομένων. Δεν πρέπει να δούμε λοιπόν την κινητικότητα θεωρητικά αλλά και τις συγκεκριμένες πτυχές της. Και επίσης, συμφωνώ με την κυρία Ρούλα, για την έλλειψη νομοθεσίας. Μας μιλούσε ατύπωση η Γενική Διεύθυνση της Αγοράς για τα λεγόμενα country desks, για τις υπηρεσίες ανά χώρα. Εγώ πιστεύω ότι η... να υπάρξει μια συζήτηση για ορισμένα θέματα. Όταν βλέπουμε παραγωγικά την κατάσταση τη KLM με τη Ryanair, θα πρέπει να υπάρξει μια πιο γρήγορη αλληλεπίδραση μεταξύ του Και ένα τελευταίο σημείο, όταν μιλάμε για την εφαρμογή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το πρόβλημα τη διαφοράς και των αθεμήτων εμπορικών πρακτικών που είναι και αυτά ένα πρόβλημα για την εσωτερική αγορά. Η κυρία Μακλάρκιν δεν μπόρεσε να είναι παρούσα και εγώ βρίσκω ότι χαιρετούμε την προσέγγιση της, χαιρετούμε την προσέγγιση της κυρίας Μπαστός. Απλώς θέλω να τονίσω ότι οι γνωμοδοτήσεις που θα έρθουν σε εμά από τις υπόλοιπε επιτροπές θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να μπορέσουμε να έχουμε μια ευρύτερη ισορροπία στην έκθεση αυτή γιατί κάποια θέματα πράγματι παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και έχουμε ενδιαφέροντα θέματα που ετέθησαν παραγωγής για τα πτυχία των φοιτητών. Κάποια από αυτά καλύπτονται από τη διαδικασία της Μπολόνια και όχι από τη δική μας διαδικασία αναγνώρισης προσόντων. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβηθούμε να επισημάνουμε τις ευθύνες των κρατών μελών όπου υπάρχουν, όπως είπε και η κυρία Μπάστος, είναι απαραίτητο η Κομισιόν να εξακολουθήσει να διατηρεί την πίεση πάνω στα κράτη-μέλη και όπως είπατε να πει στα κράτη-μέλη ότι πολλές φορές κατηγορούν την Κομισιόν οι πολίτες για την, τα προβλήματα της ενιαίας αγοράς, ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κράτη-μέλη τα οποία δημιουργούν τεχνητά και άχρηστα προσκόμματα, τα οποία δεν βοηθούν αυτή την κατάσταση. Και αυτό συνδέεται με αυτό που λέει η κυρία Ρούλα, ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν μπορούν να πάρουν το αυτοκίνητό τους από τη μία χώρα σε μια άλλη και να το εκτελονίσουν ή γιατί έχουν δυσκολία να έχουν ε, ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους και όπως τον η κυρία Γκέπχαρτ και η κυρία Ριούλε χθε, γιατί δεν μπορούν να έχουν ένα τραπεζικό λογαριασμό σε μια άλλη χώρα. Όλα αυτά λόγω επαχθών γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ακόμα και αν είχαν τα λεφτά δεν θα μπορούσαν να δείξουν τους λογαριασμούς. Τέτοια πράγματα λοιπόν νομίζω ότι μπερδεύουν τους πολίτες και συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος ε, De για την πρόσβαση σε προϊόντα στο διαδίκτυο που είναι ένα πρόβλημα ανταγωνισμού. Και χαίρομαι γιατί στην έκθεση που γίνεται για την οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου και την αναθεώρηση της εσωτερικής αγοράς από την Κομισιόν μπορεί να επαλέθουμε στα θέματα αυτά. Θέλει κάποιο άλλο να λάβει το λόγο ή θα δώσει το λόγο στην Κομισιόν. Κύριε Κουρή Ντικάμψου και κύριε Σουάπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τη συναδελφό μου, τη Ριζίνα Μπάστους, για αυτό το έργο της και ιδίως γιατί είχε την πρωτοβουλία, ε, έλαβε την πρωτοβουλία να συμπεριλάβει και το θέμα της ευκυβερνησίας, που είναι ένα κρίσιμο θέμα. Η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί. Ξέρουμε ότι το επίπεδο λειτουργίας της είναι χαμηλό. Αυτό έχει να κάνει όμως και με την νοοτροπία και την κουλτούρα που σε εθνικό επίπεδο πολλές φορές δεν είναι ιδιαίτερα θετική και εφεκτική. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε κάποια πίεση στα κράτη-μέλη, αλλά να εξασφαλίσουμε και ότι υπάρχει μια διαδικασία mainstream στα κράτη-μέλη, ώστε στα κοινοβούλια και στις εκτελεστικές εξουσίες να υπάρξουν οι απαραίτητες κινήσεις. Δεν θα ήταν υπερβολικό να ζητήσουμε να υπάρχει μια σύσταση, ώστε να υπενθυμίσουμε ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις <clears throat> θα πρέπει να λάβουν κάποια μέτρα για τα θέματα του περιβάλλοντος, ότι όλες οι κυβέρνησεις έχουν τη δυνατότητα, την ανάγκη να λάβουν υπόψη τα θέματα ισότητας των φύλων. Γιατί όμως οι κυβερνήσεις να μην ασχολούνται με τον ίδιο τρόπο που ασχολούνται με το περιβάλλον και τα θέματα φύλου, με τα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς. Ότι σε κάθε νομοθέτημα το οποίο <clears throat> ε, ε, εγκρίνεται να λάβουν υπόψη την ανάγκη να λάβουν υπόψη τους πολίτες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Αν το κάνουμε λοιπόν αυτό το πράγμα, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους πολίτες κάποιων χωρών να σκεφτούν περισσότερο για την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Κύριο Σφάπ, και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω με, αυτό που ανέφερε ο κύριος ε, Σφάπ. Έχουμε λοιπόν πολλές καλές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για την ενιαία αγορά. Έχουμε προσπαθήσει, έχει προσπαθήσει η κυρία Ρεζίνα Μπάστος να περιλάβει αυτά τα 20 στοιχεία, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα ότι τα κράτη-μέλη εμποδίζουν σε πολλά σημεία την ενιαία αγορά, όπως είδαμε και με το δίκαιο των συμβάσεων. Το αν χρειάζεται τώρα μια κεντρική υπηρεσία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά τα κράτη-μέλη έχουν τα στοιχεία τα οποία δεν δίδουν σε άλλου. Δεν είναι σωστό να θεωρεί κανεί ότι αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη είναι σωστό και αυτό που κάνει η Ευρώπη είναι λαθασμένο. Χρειάζεται μια ισορροπία, δεν είναι το μόνο σημείο στο οποίο χρειάζεται ισορροπία. όπω είπε και ο συνάδελφο De Jong, δεν θα πρέπει να τα κάνουμε όλα πάσα στην Ευρώπη πρέπει και αυτό να το καταλάβουν οι πολίτες ότι χρειάζεται μια ισορροπία και θέλω εγώ να επενέσω την κυρία Μπάστος. Είδα το ίδιο το κείμενο αυτό και έχω συζητήσει με τις περιφερειακές αρχές και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει στο να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς και οι πολίτες. Δεν πρέπει να έχουμε μονάχα τα προβλήματα, να βλέπουμε μόνο τα προβλήματα για την Ευρώπη. Θα πρέπει να τονίσουμε και τα θετικά της στοιχεία. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Απλώ να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο τη Επιτροπή, κυρία Πανχόφεν. Και μετά η κυρία Μπαστό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, ευχαριστούμε ιδιαίτερω την κυρία Μπαστό και την Επιτροπή σα που ετοιμάζει την έκθεση αυτή. Τη βρίσκουμε πολύ επικοδομητική. Μα ικανοποιεί ιδιαίτερω και η όλη συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα, διότι και εμείς θα συμφωνήσουμε με την έκκλησή σα για περισσότερο σφαιρική προσέγγιση στην εσωτερική αγορά. Και να φροντίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε σε καθημερινό επίπεδο να λειτουργεί η εσωτερική αγορά. Να δούμε τι εμείς μπορούμε να κάνουμε, αλλά και τι θα έπρεπε να κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτά ήθελα να πω. Λίγο πολύ. Σα ευχαριστώ. Συμφωνούμε με το πνεύμα που περιγράψατε εδώ. Uh, well, θα δείτε τις νομοδοτήσεις και των υπολείπων επιτροπών. Ζητήσαμε να είναι φάνταστες τις λύσεις που θα προτείνουν και να συμπληρώσουν την έκθεση της κυρίας Μπαστός όσο καλύτερα γίνεται. Θέλετε να συμπληρώσετε εσείς κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα να συνοψίσω. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνεισέφεραν σε αυτή τη συζήτηση. Μου φαίνεται δεν υπάρχουν αποκλήσεις απόψεων στα μεγάλα ζητήματα Θέλουμε ουσιαστικά να κατακτήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και να τους πείσουμε για τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνη σήμερα και αυτή ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να αναζητήσουμε την κατάλληλη λύση, όπως είπε σωστά ο Πρόεδρος και εγώ προσυπογράφω όλο χερό αυτό που είπατε, δεν πρέπει να φοβόμαστε να κάνουμε συστάσει προ τα κάτι μέλη. Αυτή η έκθεση είναι ακριβώ το η τέλεια ευκαιρία για να κάνουμε συστάσεις προς τα κάτι μέλη στην κατεύθυνση του να είναι περισσότερο πειθαρχημένοι και να προβάλλουν τις αρετές και τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό είμαι ανεπιφύλακτη. Και σωστά το είπε και ο συνάδελφος Δεκάμπους ότι θα πρέπει να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε ευθυγράμμιση, ευθυγράμμιση της νομοθεσίας που πρόκειται να υιοθετήσουν στο μέλλον και η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί ως προς τον αντίκτυπό της. Για τα ωφέλη και τις συνέπειες που θα έχει στο επίπεδο της εσωτερικής αγοράς, ως προς τις ε, νημερωτικές εκστατείες. Είναι θεμελιώδου σημασίας αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η διάδοση πληροφοριών, η καλή πληροφόρηση και τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς πρέπει να φτάσουν πια στους πολίτες, ώστε να μπορεί να λειτουργεί η εσωτερική αγορά αξιοποιώντα όλα αυτά τα πλεονεκτήματα το ίδιο και τι επιχειρήσει. Είναι σημαντικέ αυτέ οι εκστρατείε σε αλληλεπίδραση με του πολίτε, όπω είπε και ο συνάδελφο Νταγιό, πολύ σημαντικό. Και εδώ θέλουμε και την δέσμευση, τη συμμετοχή των κατώμελών. Αυτό ακριβώ θα περάσει μέσα από τι συστάσει για να αντιμετωπιστεί το θέμα των κενών που εντοπίσαμε η συμμετοχή των κρατών μελών. Τώρα, το ζήτημα του νομοθετικού επίπεδου, εάν θα πρέπει αυτά να επιλύονται σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. Η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες επειδή ε, έτσι βλέπουν και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δυνατότητα δηλαδή να νομοθετεί σε τέτοια ζητήματα, σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ακόμη και εάν ε, θέλουμε να, είμαστε, να υπάρχει εγκύτητα στην νομοθεσία και είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό, υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Να ολοκληρώσω λοιπόν, ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους για τη συμβολή τους και πραγματικά νομίζω ότι ολοκληρώνοντα και αξιολογώντα τι νομοθεσίες και των υπολείπων επιτροπών, θα έχουμε πραγματικά μια έκθεση που θα συμπεριλαμβάνει τα σημαντικά μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε προς τα κράτη-μέλη. Το ίδιο και για το Συμβούλιο και την Επιτροπή από την πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. απλώ να επιβεβαιώσω ότι οι προθεσμοί για τι τροπολογίε είναι η 12η Απριλίου στι 12 το μεσημέρι και θα συνεδριάσουμε στις 8 Μαΐου για την εξέταση των τροπολογιών και να δούμε και τι γνωμοδοτήσει των άλλων επιτροπών συγχρόνω. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, κύριε Μπαστό. Ήταν το τελευταίο θέμα. Ευχαριστώ του διερμηνεί όπω πάντα, που μα δώσαν λίγο πρόσθετο χρόνο, δωρεάν κιόλα. Επόμενη συνεδρίαση είναι 5η 12 Απριλίου, είναι νέα ημερομηνία για την ε, τμήμα των νέων μέτρων. Θα έχουμε λοιπόν στις 12 Απριλίου 9 με 12.30 και στη συνέχεια 25 και 26 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Τέρμα. AUTHORWAVE